Αρχίζει η συνεδρίαση. Καλημέρα σας. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού. Η πρώτη συζήτηση αφορά τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών ελευθεριών στην Μπουργκίνα Φάσο. Να σας υπενθυμίσω και πάλι ότι μπορείτε να ζητήσετε το λόγο για να μιλήσετε με catch the eye ή με γαλάζια κάρτα χρησιμοποιώντας τόσο το συνήθι τρόπο εγγραφής όσο και το νέο σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής. Οι σχετικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στην είσοδο του ημικυκλίου. Από τους συντάκτες το λόγο έχει πρώτη η κυρία Κάνκο για ένα λεπτό. Η καρδιά μου ματώνει. Η πατρίδα μου, Μπουρκίνα φάσω. κάποτε ήταν κοσμικό κράτος και τώρα στενάζει από το τρόμο της Ισλαμικής ε, και της βίας. Είδαμε ε, πρώτα που έσπηραν στη Συρία το θάνατο και τον τρόμο και τώρα έχουν επεκταθεί και μέχρι την Αφρική με την τρομακτική ε, τους ιδεολογία του θανάτου. Επιτίθενται και σε εκκλησίες και σε ε, τεμένοι. Αυτό που θέλουν είναι να καταστρέψουν την κοινωνία τους νοιάζει να καταστρέψουν τους χώρους όπου συγκεντρώνεται ο κόσμος για τη λατρεία, για την αγάπη, για να ψέλνει, για να προσεύχεται. Υπάρχουν γεωπολιτικές συνέπειες τεράστιες, κυρίως για την Ευρώπη. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, αλλά να μην ξεχνάμε και ε, ε, τα τρομοκρατικά χτυπήματα στην καρδιά της Ένωσης. Γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίζει να υποστηρίζει τις χώρες Σαχέλ για να εγγυηθεί την ασφάλεια στην περιοχή, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνεργασία στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρική. θα πρέπει να απαντήσουμε με ανάπτυξη και ευημερία, να μην αφήσουμε στη μοίρα τη την Πουρκίνα Φάσο και το ε, Σαχέλ. Αλλιώ θα υπάρξει χάο και πολύ γρήγορα θα τα βρούμε μπροστά μας στην Ευρώπη. Μην ξεχνάτε ότι ήταν κοσμικό κράτος η Μπουρκίνα Φάσο. Το, το λόγο έχει κυρία για ένα λεπτό. No one should be subjected to violence because of their religion Κανεί δεν θα πρέπει να εφίσταται την ε, βία λογοθρησκείας ή για άλλο χαρακτηριστικό εθνοτικής καταγωγής, εξωτερικών προτιμήσεων, πολιτικών πεπιθήσεων, κανείς και ποτέ. Δυστυχώς όμως έχουμε 750 νεκρούς φέτος χιλιάδες ε, τους εκτοπισμένους ε, φτάνουμε σε ανθρωπιστική τραγωδία αλλά η χώρα έχει μακρά ιστορία ανεκτικότητας θρησκευτική και πρέπει να αποτίσουμε φοροτιμή σε όλου αυτούς τους ταραλέους οι οποίοι με βάση εκείνη την παράδοση προσπαθούν να αντισταθούν σε αυτές τις ε, συγκρούσεις γιατί οι ένοπλε διαφορέ, οι ένοπλες ε, αναμετρήσει δεν ε, λύνουν τίποτε, έχουμε όλο ένα και περισσότερο τσοσβαστικοποίηση και θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, οι διοικητικές αρχές να κάνουν το ίδιο, να υπάρχει αξιοπρέπεια ε, και ανάπτυξη και ελπίδα. Πάρα πολλές πιέσεις υπάρχουν, κλιματική αλλαγή, έχει φυγεί το βιωτικό επίπεδο της χώρας, αλλά και η ΚΑΠ ε, οφείλεται, διότι έχει πλήξει με τα μέτρα της την τοπική γαλακτοβιομηχανία. αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια συνεκτική πολιτική, θα πρέπει να υποστηρίξουμε όλους όσους ε, αντιτάσσονται στον εξτρεμισμό και να τους βοηθήσουμε να επαναφέρουν τη χώρα στην ειρήνη και το διάλογο. Κυρία Αρένα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Μπουρκίνα Φάσο είναι μια χώρα κοσμική. Η πρώτη χώρα τη Δυτική Αφρική που δημιούργησε την αδερφοσύνη των πιστών, όπου προεδρεύει και συμπροεδρεύει από το 1972 ε, ομάδα χριστιανών και μουσουλμάνων. Η Μπουρκίνα Φάσο, λοιπόν, έχει μεγάλη παράδοση διαθρησκιακού διαλόγου. Δυστυχώ, από το 2015, η Μπουρκίνα Φάσο, όπω και όλε οι χώρε του Σαχέλ, έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά φαινόμενα βία. Ε, οι οποίε απειλούν την κοινωνία των πολιτών λόγω των τζιχαντιστών και των ένοπλων ομάδων και στοχεύουν όλες τις ε, μετριοπαθεί θρησκευτικέ ομάδες. Ε, έτσι, η βάση της χώρας αυτής, η βάση διαλόγου και ανοιχτής διάθεσης απειλείται. Προσπαθούν να δημιουργήσουν άνομες περιοχές στην περιοχή του Σαχέλ. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα γενεσιοργά αίτια, τη φτώχεια, την αδυναμία του κρατικού συστήματος και τη διαφθορά που μαστίζει την χώρα. Η ασφάλεια θα πρέπει να, να υπάρξει στην περιοχή αυτή ώστε να ενισχύσουμε την προστασία του Σαχέλ στην όλη μας δράση. Και θα πρέπει να υπάρξει κατεπίγουσα προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας για την περιοχή αυτή, διότι πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι σήμερα υποφέρουν από πείνα. Δεν μπορούμε με μόνη δικαιολογία την ασφάλεια να ξεχνάμε τη φτώχεια και την ανθρωπιστική βοήθεια που είναι πρωταρχική σημασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Βιλανόεβα Ρουή για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην περιοχή του Σαχίλ έχουμε μια ανθρωπιστική κρίση πάρα πολύ σοβαρή. Τρομοκρατικές ενέργειες και έχουμε ε, ένδια και επίσης ε, έχουμε περισσότερους ε, νεκρούς το 19 προς το 18 και το πρόβλημα είναι το πώς θα υπάρχει ασφάλεια με την αμυντική έννοια να βελτιωθεί η ασφάλεια και ένα δεύτερο στοιχείο είναι το ότι οι Αφρικανοί χρησιμοποιούν τόσα χέρια να φτάσουν στην Ευρώπη. Έχουμε σταματήσει την ε, πολιτική ασφάλειας και ανθρωπινών δικαιωμάτων η ασφάλεια δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το πώς οι μετανάστες έρχονται, αλλά θα πρέπει να, είναι, να έχει πνεύμα δικαιοσύνη. Μεταπικιακή είναι η πολιτική μας, αλλά δεν χρειάζεται να βοηθήσουμε τα αγροδιατροφικά για να μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι εκεί στην Ήπεθρο, να οικοδομηθεί ασφάλεια και ειρήνη. Δημοκρατία ενισχύοντας την κοινωνία των πολιτών και τα αιτήματα αυτής και όχι τα οικονομικά συμφέροντα που πολλά από αυτά είναι ευρωπαϊκών πηγών και αυτά επιδεινώνουν την κατάσταση. Λόγο έχει ο κύριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Η κατάσταση στα κράτη του Σαχέλ είναι πραγματικά ζωφερή αυτή τη στιγμή και στην Πορκίνα Φάσο. Οι χώρες του Σαχέλ θα πρέπει να ειδωθούν συνολικά. Είναι και το Μαλί και ο Νίγηρας και τα λοιπά. Δεν είναι μόνο η Πουρκίνα Φάσο. Ε, και ακούσαμε ότι η χώρα αυτή ήταν κοσμική. Ε, συμβίωναν ειρηνικά οι θρησκείες παλιά. Δεν ισχύει αυτό σήμερα. Δεν είχε σημασία ε, σε ποια θρησκεία ανήκε στο παρελθόν. Σήμερα αυτό έχει καταργηθεί δεν κυνηγάνε μόνο τους χριστιανούς οι αλλά και τους μετριοπαθείς μουσουλμάνους. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια κατάσταση και ε, μια κουλτούρα με μεγάλη δυσπιστία, με μεγάλα προβλήματα ε, στο διαθρησκιακό διάλογο. Και γι' αυτό πιστεύω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούμε, να ενισχύσουμε περισσότερο αυτή την περιφέρεια, να δώσουμε μια προοπτική στον κόσμο για να μην ριζοσπαστικοποιούνται οι ανθρωπικοί, αλλά χρειάζεται και στρατιωτική υποστήριξη. Μόλι είπε η συνάδελφο ότι η ασφάλεια δεν εξαρτάται από το πόσου ε, στρατιώτε στέλνουμε, ε, λοιπόν εξαρτάται και από αυτό. Και ω Ευρωπαίοι θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγαλύτερη παρουσία και ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριο Χολβίνη για ένα λεπτό. Ε, αξιότιμοι συνάδελφοι ε, συζητούμε σήμερα επιτέλου επιτέλους αυτό το θέμα. Ε, καταφέραμε ε, να ασχοληθούμε με την να Φάσο. Έχω συνυπογράψει αυτό το αίτημα και είναι πάρα πολύ καλό που ε, έφτασε η συζήτηση στην Ολομέλεια. Χρειάζεται βοήθεια ο κόσμος εκεί. Εδώ και μήνες διαβάζουμε ότι υπάρχει τρομοκρατική βία που πλήττει τη χώρα. Τζιχαντιστές επιτίθενται σε χριστιανούς και όχι μόνο και σε μετριοπαθείς μουσουλμάνους. Ε, είναι μακρά η παράδοση συμβίωσης των θρησκειών εκεί στη χώρα, η ειρηνική συμβίωση η οποία καταστρέφεται. Και τώρα επικρατεί χάος. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις από την ε, Ουγγαρία. Έχουμε ένα πρόγραμμα, η Ουγγαρία βοηθάει, Hungary Helps, κατά της ε, βίας αυτής και κατά των φαινομένων στην Πουρκίνα Φάσο. Μα εξήγησε ο γραμματέα τη οργάνωση αυτή τι συμβαίνει, πώ έχουν τα πράγματα επί τόπου και γνωρίζουμε ότι η κατάσταση αφορά όλη τη χώρα και είναι 600.000 οι εσωτερικοί πρόσφυγες και εκτοπισμένοι.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 ε, και στην Πορκίνα Φάσο επικρατεί χάος. Εκεί μουσουλμάνοι και χριστιανοί ζούσαν ειρηνικά. με που πριν από λίγα χρόνια είχαμε φωνικές επιθέσεις ε, με ομάδες που συνδέονται με την Αλκάιντα και τον Ούσρατ Αλ-Ισλάμ. Τρομοκρατικά χτυπήματα κατά χριστιανών και μετριοπαθών μουσουλμάνων σε ένα, Σαββατο... ένα Σαββατοκυριακό επιτέθηκαν ε, και σε εκκλησίες και σε σχολεία και ε, διώκουν πολλούς χριστιανούς οι οποίοι ε, είναι σε φυγή. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Και τα προβλήματα δεν είναι μόνο από τα τρομοκρατικά χτυπήματα, αλλά και από την ξηρασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να βοηθάει αυτή τη χώρα, να εντείνει την παρουσία της και την βοήθειά της σε όλη την περιοχή. Θα πρέπει απερίφραστα να καταδικάζουμε αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις και ή δυνατόν να τις αποτρέπουμε. Για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών το λόγο έχει η κυρία Γκίλ για ένα λεπτό. Thank you, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπατε εκπρόσωπε, η κατάσταση στην Πορκίνα Φάσο διαρκώ υποβαθμίζεται μέσα στα χρόνια. Και είναι σημαντικό να κοιτάξουμε την κατάσταση σφαιρικά. Όχι να επικεντρωνόμαστε σε μία ομάδα ή μία χώρα. Αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει πάνω απ' όλο είναι ότι η περιοχή του Σαχέλ έχει γίνει, όπως ήδη ακούσαμε, ε, μια αιστεία ανάπτυξης για το ISIS, που ε, εκμεταλλεύεται την αστάθεια μια ε, περιοχή του κόσμου που έχει τη χειρότερη διακυβέρνηση. Ε, η στρατηγική που θα αναπτύξουμε είναι σημαντική για την Δυτική Αφρική. Πρέπει να υποστηρίξουμε τι χώρε αυτέ, διότι οι ένοπλε δυνάμει ε, δεν έχουν αρκετό δυναμικό και οι στρατηγικέ των ίδιων των χωρών δεν μπορούν να διατηρήσουν τη σταθερότητα. Η καταπολέμηση, η πολιτική μάλλον τη εκτέλεση των υπόπτων απλώ υποδαβλίζει την διένεξη και ουσιαστικά ε, δίνει περισσότερα επιχειρήματα στους ε, εξεγερμένους. Πώς θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να οργανώσει τις ε, έρευνες με κοινέ δυνάμεις και τι θα κάνει γι' αυτό. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στα θέματα συμμόρφωσης με τα, δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα από όλες τις περιοχές τη περιοχή. Ομάδα Renew, το λόγο έχει η κυρία Ράμος. Για ένα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριε, είπατε εκπρόσωπε, η Μπουρκίνα Φάσο είναι μεταξύ των 10 φτωχότερων κρατών του κόσμου και από το 2015 ζει μια ανίποτη και άνευ προηγουμένου βία. Ε, στο πρώτο εξάμεινο του 19 ήταν πάνω από 300 οι τρομοκρατικές επιθέσεις και οι τρομοκρατικές ένοπλες τζιχαντιστικές ομάδες έχουν μετατρέψει τη ζώνη αυτή σε ζώνη στρατολόγησης νέων και φέτος επιτίθενται σε σχολεία, τζαμιά, εκκλησίες. Αυτό είναι το ε, σχήμα. Και πάνω από μισό εκατομμύριο είναι εσωτερικά εκτοπιστέντες που έρχονται να προσθεθούν και ε, στους εκτοπισμένους από το Μαλί. Τι θα γίνει τώρα. Το 80% του πληθυσμού εξαρτάται από τη βοήθεια στην ε, γεωργία για να επιβιώσει και ο υποσυτισμός έχει χτυπήσει κόκκινο. Γι' αυτό το Σαχέλ χρειάζεται στρατηγική καταπολέμηση τη τρομοκρατία, ε, στρατηγική ειρήνη και σταθερότητα και ασφάλεια. Αλλά η Μπουρκίνα σήμερα χρειάζεται και πήγουσα επισητιστική βοήθεια και ε, στην ανάπτυξη. Για την ομάδα των Πρασίνων, το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριο Σατούρη. Το ψήφισμα αυτό διαγράφει το σχεδιαγραφεί μάλλον το δύσκολο τοπίο της Μπουρκίνα Φάσο. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο διαθρησκιακός διάλογος θα πρέπει να αποτελεί πυλώνα συνέπραξη στην ε, Μπουρκίνα Φάσο. Η θρησκεία και η δυνατότητα εθνικής ενότητας υπάρχει ακόμα. Εδώ λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια πολιτική κρίση. Κρίση ε, στις χώρες ε, γενικότερα εκεί. Και αυτό έχει να κάνει με την υπερθέμανση του πλανήτη. Η Μπουρκίνα Φάσο μάχεται ώστε η ακραία φτώχεια, ο λοιμό, να μην γίνει εστία ανάπτυξη για τον τζιχαντισμό. Οι χώρες της Ευρώπης έχουν εδώ να ευθύνη και η δράση μας θα πρέπει να γίνει αντιληπτή από τον πληθυσμό, πληθυσμό πράγμα που δεν συμβαίνει ω τώρα. Μέχρι τώρα έχουμε αποτύχει και θα πρέπει με τις ε, προσπάθειες που έχουμε κάνει ως τώρα να φροντίσουμε να τις εντείνουμε. Η Γαλλία και η υπόλοιπη διεθνής κοινότητα, οι ευρωπαϊκές χώρες, να βοηθήσουν την κοινότητα των χωρών του Σαχέλ. Πρέπει να κάνουμε ένα ειλικρινή και έντιμο απολογισμό, να αντλήσουμε τα διδάγματα από μακρά ιστορία αποτυχιών. Μόνο με τους πληθυσμούς, τους πολίτες στο πλευρό μας, μπορούμε να επανοικοδομήσουμε την σταθερότητα στις χώρες αυτές. Σας ευχαριστώ για την ομάδα ταυτότητας και δημοκρατίας. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ και λίγο χρόνο γίνεται δίωξη των χριστιανών, αλλά όχι μόνο αυτών. Έχουμε πάνω από 12 ομάδες διχαντιστών που έχουν σχέση με την Αλκάιντα και από το 12 με το 2015 ε, έχουν προκαλέσει 750 ανθρωποκτονίες, έχουν προκαλέσει επίσης την έξοδο ανθρώπων από τα χωριά τους, εκτόπιση και έχουμε 74 χριστιανούς επίσης, τρεις ιερείς και ε, η τελευταία επίθεση έγινε την ε, Κυριακή σε κάποια χριστιανική γιορτή μέσα σε μια εκκλησία ε, σκότωσαν ανήλικους για τον ίδιο τον ιερέα που έκανε τη λειτουργία έχει γίνει επομένως τώρα ένα τόπος μαρτυρίου για τις μειονότητες θα πρέπει το Κοινοβούλιο να λάβει υπόψη ότι δεν είναι μόνο μια πλούσια χώρα, αλλά είναι και ευάλωτη χώρα και θα πρέπει αναλόγως να αναλάβουμε δράση και θα πρέπει κάτι να κάνουμε για αυτούς τους χριστιανούς που παίζουν τη ζωή τους για την ε, ε, πίστη τους τώρα που κοντά τα Χριστούγεννα και θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη ότι αυτοί οι άνθρωποι κηρύσουν την πίστη τους και γι' αυτό και χάνουν τη ζωή τους. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Ρούισεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η ε, ε, ακραία ε, Ισλαμιστική βία έχει αλλάξει την Μπουρκίνα Φάσο. Μια χώρα που ήταν τόσο φιλιρινική, με ανεκτικότητα θρησκευτική, έχει γίνει τώρα σφίγγοφολιά των εξτρεμιστών. Η χριστιανική μειονότητα πλήττεται σφοδρά. Μόνο το 2019 πάνω από 60 χριστιανοί δολοφονήθηκαν από στοχευμένες επιθέσεις. Κλείνουν εκκλησίες και διώκονται οι χριστιανοί από τα χωριά τους. Ανησυχώ βαθύτατα. Πολύ δε περισσότερο που η βία δεν περιορίζεται στην Πορκίνα Φάσο, αλλά αυξάνεται σε όλη την περιοχή του Σαχέλ. Χρειάζεται οπωσδήποτε επιγόντως διεθνής δράση. Καλό την Ευρωπαϊκή Ένωση να κοιτάξει την κατάσταση των χριστιανών στην περιοχή ε, και να τη συμπεριλάβει στην κοινή πολιτική ασφαλείας και στη νέα στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής. Δεν μπορεί να εξαφανιστεί η χριστιανική παρουσία στην Πορκίνα Φάσο και στην περιοχή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Το λόγο έχει η κυρία Μπενσουμέα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δυστυχώς, η περίπτωση που σήμερα καταδικάσουμε η επίθεση σε χριστιανικό ναό στην Μπορκίνα Φάσο δεν είναι απομονωμένη, η μεμονωμένη περίπτωση. Ε, τα τελευταία χρόνια ζούμε μια πραγματική χριστιανική δίωξη. Διωγμούς ζουν οι χριστιανοί. Όχι μόνο στην Μπορκίνα Φάσο, Νιγηρία, Αφγανιστάν, Σομαλία, Σρι και πάει λέγοντας. Ε, αυτή η δίωξη για θρησκευτικούς λόγους προέρχεται από Ισλαμιστές, τρομοκράτες κατά χριστιανών που τους ε, δολοφονούν ψυχρό επειδή ε, λατρεύουν το Θεό τους. Ε, ανατριχιαστικά τα στοιχεία της Open Doors το 2018 πάνω από 4.000 χριστιανοί δολοφονήθηκαν επειδή είχαν πάει στην εκκλησία. 3.125 ε, συνελήφθησαν και πάρα πολλές εκκλησίες ε, καταστρέφονται. Αυτό είναι επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ζήση, των αξιών μας, του τρόπου ζωής μας και τελικά επιθέσεις κατά της ίδιας μας ελευθερίας και δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Τζόουνς για ένα λεπτό. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Άλλοι συναδελφοί μίλησαν για την κατάσταση στην Πουρκίνα Φάσο ε, που είναι γνωστή ότι ήταν χώρα με ανεκτικότητα σε διαφορετικές κουλτούρες και θρησκείες. Μπράβο στους ε, ε, συναδελφούς που τα αναφέρανε. Πρόκειται για κάποιες επιθέσεις, αποτρόπες, αλλά θα πρέπει να προβλημαστούμε στο πλαίσιο της γενικότερης θεματολογίας προβληματικής και συλληπιτήρια προς τις οικογένειες όσων ε, έχουν φωνευθεί, ε, όσων ε, περνάνε όλα αυτά λόγω αυτών των επιθέσεων. Και δεν μιλώ μόνο για την Πουργία Φάζο, για όλο τον κόσμο σας λέω. Και από ό,τι γνωρίζω, η βία είναι ένα μικρόβιο, αρρώστια που θίγει χώρες, δημοκρατίες, τη ζωή μας, την καρδιά μας, οπότε θα πρέπει να την φρενάρουμε με κάθε τίμημα. Και τι εννοώ, Νομίζω ότι καμία χώρα δεν είναι θωρακισμένη από τέτοιε επιθέσει. Θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε, τι στρατηγική θα έχουμε Ευρώπη, Αφρική, πώ θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη, συνεργασία και φιλία. Και οπωσδήποτε χρηματοδότηση, θετικέ ενέργειε και όχι αρνητικέ, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ο κόσμο είναι ένα και δεν χωρεί διχασμού και διαρρήσει. η σωρία ε, παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιθέσεων στην Πουρκίνα Φάσο πραγματικά μας αφήνει άφωνο. Στρατιωτικές και ένοπλες δυνάμεις ε, στρέφονται κατά εκκλησιών, σχολείων. Ε, η κατάσταση επιδεινώνεται διαρκώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στοχεύσει τη βοήθειά τη ώστε να μπορέσει να ενισχύσει την ασφάλεια στην ε, περιοχή και κυρίω τι δημοκρατικέ δυνάμει τη χώρα. Πρέπει να επενδύσουμε μακροπρόθεσμα σε ε, σχολέ εκπαίδευση για την αστυνομία, την χωροφυλακή, τον στρατό. Θα πρέπει οι χώρε αυτέ να ξεπεράσουν αυτέ τι αδυναμίε και να είμαστε κι εμεί παρόντε στην πράξη για να δούμε τι εκπαίδευση παρέχουμε. Πρέπει όμω και οι αρχέ τη Μπουρκίνα Φάσο να μα πούν πώ θα επανακατακτήσουν την και τι στήριξη θέλουν από εμά. Στήριξη στα κριτική, αλλά και ταυτόχρονα μια στήριξη για τι ε, ε, διοικητικέ δυνάμει εσωτερικώ, για τα τελωνία και τη δικαιοσύνη. Δεν έχουμε πια χρόνο. Χρειάζεται ευρωπαϊκή στρατηγική για το Σαχέλ, ώστε να μπορέσουμε να αγωνιστούμε μαζί με του ε, κατοίκου εκεί. Έχουμε όλα τα όπλα στη διάθεσή μα, όλα τα μέσα, αλλά πρέπει καλύτερα να συντονιστούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση που είναι σημαντική για την ασφάλεια στη Σαχέλ. Είναι μια πρόκληση για την Αφρική, αλλά είναι και για μα. Σα ευχαριστώ. Το λόγο έχει κυρία Μπίλτ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μισό εκατομμύριο εκτοπισμένοι. Δύο χιλιάδες σχολεία σχεδόν έχουν κλείσει και είναι και στόχοι καμιά φορά. Γιατί επειδή εκεί γίνεται μάθημα στα γαλλικά. Ε, ε, είναι ένοχοι οι σιωποί ε, της Δύσης. Βλέπουμε στις αρχές ε, του μήνα επίθεση σε προτεσταντικό ναό ε, σε ανατολική χώρα με απολογισμό 14 θύματα. Έτσι συχνά ε, ε, ξεφτίζει το κράτος που ήταν εγγύηση σταθερότητα στη Δυτική Αφρική. Και έτσι ολοκληρώνεται και ανάφλεξη του Σαχέλ από μια σύγκρουση που στην αρχή ήταν περιορισμένη στο Βόρειο Μαλί. Ε, πώς να απορεί κανείς όταν ξέρουμε ότι μόνο 4.500 Γάλλοι στρατιώτες είναι χαμένοι σε μια τεράστια ήπειρο στο Σαχέλ. Ενώ ε, στο Μαλί ε, δεν ε, υπάρχει δυνατότητα αντίδραση. Ακούω του συναδέλφου, κυρία Λουαζό, όλοι συμφωνούμε. Ωστόσο, Ωραία τα λέμε εδώ στη βολή του Κοινοβουλίου, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα εάν δεν καταλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι διακυβεύεται εκεί. Το μέλλον είναι κρίσιμο και για το χριστιανισμό και για την ίδια την Ευρώπη. Σημειώστε το αυτό σήμερα που είναι και Χριστούγεννα σε λίγο. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Πορέμπα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει να καταδικάσουμε περίπτωση αυτές τις επιθέσεις και θα πρέπει να τοποθετηθούμε με ελληνική για τον κόσμο εκεί. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αναλογιστούμε το τι μπορούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, να επανέλθει σταθερότητα στη χώρα και θα πρέπει η γενικότερη περιφέρεια, η γενικότερη περιοχή να γνωρίσετε σταθερότητα. Όμω έχουμε επιθέσει ιδίω κατά χριστιανών. Αυτό γίνεται από ριζοσπαστικοποιημένου Ισλαμιστέ, έχουν σχέση με την ε, είναι πολλές οι ζωές που έχουν χαθεί. Τώρα πρόσφατα επιτέθηκαν σε κάποια εκκλησία όπου είχαμε πολλές δεκάδες πιστών ε, μεταξύ των οποίων και παιδιά που πυροβολήθηκαν με τα πολυβόλα. Επομένως θα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες ενέργειες για να ξαναγυρίσει σταθερότητα στη χώρα και βέβαια ε, ο ύπατος εκπρόσωπος έχει πολλά να κάνει σε αυτό το μέτωπο. Χρειάζεται μια καινούργια στρατηγική, ανθρωπιστική αρρωγή και συγκεκριμένε πρωτοβουλίε. Το λόγο έχει ο κύριο Χέτμαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Την 1η Δεκεμβρίου είχαμε αυτήν την ένοπλη επίθεση κατά της Εκκλησίας όπου 14 εφωνεύθησαν και πολλοί τραυματίστηκαν. Το 19 οι τζιχαντιστές σκότωσαν 40 χριστιανούς και όλό ένα και περισσότεροι είναι η βία στη χώρα. Μιλούμε για εκατοντάδες χιλιάδων που εκτοπίστηκαν. Εκατοντάδες έχουν χάσει τη ζωή τους και τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται, κλείνουν οι εκκλησίες, οπότε θα πρέπει η χώρα να αναλάβει πιο αποφασιστική δράση, να προστατεύσει τις θρησκευτικές Μειοψηφίε να καταπολεμήσει τη ρουσμαστικοποίηση. Έχει πολλά προβλήματα η χώρα. Ε, είναι μία από τις δέκα πιο φτωχέ χώρες στον κόσμο. Μαστίζεται από εμφυλίους πολέμου και η κυβέρνηση για αυτό δεν μπορεί μόνη τη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, άρα θα πρέπει να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση, με την ομάδα χωρών Σαχέλ. Όλοι οι εμπλεκόμενοι να οδηγήσουν τη χώρα στην ειρήνη, στη σταθερότητα, να συνεχίσουμε την ανθρωπιστική μας πρωτοβουλία. Το λόγο έχει ένα λεπτό ο κύριος Κούς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εμείς θα υπερψηφίσουμε το ψήφισμα. Ωστόσο, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα πολιτικά μέτρα δεν λύνουν το βασικό πρόβλημα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διωγμών των χριστιανών. Και μόνο ο αριθμός των χριστιανών που διώκονται έχει Είναι πάνω από 200 εκατομμύρια. Το τελευταίο Σαββατοκυριακό ε, σκότωσαν Ισλαμιστές στο Κονγκό 33 ανθρώπους. Αυτή είναι η απάντησή μας σε αυτό το φωνικό μίσος. Οι χριστιανοί θέλουν να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Ιησού. Αγαπάτε αλλήλους, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Και είπε στους Αποστόλους ο Ιησούς, «Ε, αφού με δίωξαν εμένα θα διώξουν και εσάς. Όμως η αγάπη μπορεί να είναι πραγματικά η απάντηση. Μπορεί. Γιατί και ο ίδιος ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο που του έδωσε το γιο του. Και αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα των Χριστουγέννων. Μόνο αυτό μπορεί να μας σώσει και να μας βοηθήσει στη σημερινή αβεβαιότητα. Γι' αυτό μας εύχομαι σε όλους χαρούμενα, ευλογημένα Χριστούγεννα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογο των εγγεγραμμένων ομιλητών. Προχωρούμε στη διαδικασία του Catch the Έχω δεχτεί τέσσερα αιτήματα και τα τέσσερα γίνονται αποδεκτά. Το λόγο έχει ο κύριος Πόσπισιλ για ένα λεπτό. ευχαριστώ πολύ. Άκουσα όλη τη συζήτηση. Οι εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι η νέα πολιτική και ε, τι ε, πρέπει να κάνουμε απέναντι σε αυτή τη συγχυσμένη χώρα. Αυτή η χώρα στο παρελθόν ήταν πάρα πολύ φιρινική με ε, ανεκτικότητα για τις θρησκείες. Τα πράγματα είναι πολύ ζωφερά. Ε, το θέμα είναι πώς θα βοηθήσουμε τώρα και τι ε, μπορούμε να κάνουμε για να βοηθηθεί η διακυβέρνηση η της χώρας δεν μπορεί να ελέγξει αυτές τις επιθέσεις. Το περασμένο εξάμεινο είχαμε δεκάδες επιθέσεις κατά των αμάχων και η κυβέρνηση δεν τα βγάζει πέρα. Τι θα κάνουμε. Θα συζητήσουμε τι πρότιθα να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το λόγο έχει η κυρία Γκραπίνη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το είπαν ήδη οι συνάδελφοι. Ε, σε λίγο έχουμε γιορτινές μέρες και δεν μπορούμε να ανεχόμαστε μια κατάσταση όπως αυτή της Μπουρκίνα Φάσο με βία, βαναυσότητα, δολοφονίες. Ε, θα πρέπει να περάσει από το ψήφισμα για να γίνει κάτι. Ε, θα πρέπει να δούμε το γεγονός ότι για την ώρα η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αξιοποιείται σωστά. Πρέπει να υπάρχει και μια πραγματική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή αυτή. Ε, μιλάμε για ανθρώπινα όντα. Χρειάζονται πραγματικά ε, χειροπιαστά μέτρα για την ε, ασφάλεια. Η ζωή των ανθρώπων δεν έχει τιμή και και από τη μια έχουμε ακραία φτώχεια, ο κόσμος ε, πεθαίνει ε, και από την άλλη έχουμε τα φαινόμενα βίας, τις ένοπλες επιθέσεις. Αυτές οι επιθέσεις λοιπόν, οι τρομοκρατικές ενέργειες, ε, είναι θέμα που αφορούσε και την, τον ΟΗΕ. Η στρατηγική του ΟΗΕ όμως και η δική πρέπει να συντονιστούν. Πρέπει να προβλέψουμε τα κατάλληλα μέτρα, διότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Γουάλλας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Μπουρκίνα Φάσο και το Σαχέλ είναι περιοχές προβληματικές τη σημερινή ημέρα. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θετικό μπορεί να κάνει. Θα πρέπει να αλλάξει στρατηγική για αυτή την ε, περιοχή θα πρέπει κάτι να κάνουμε για τις αιτίε της αστάθειας. Την αλλαγή του κλίματος, ε, βοήθεια προς την οικονομία, να σταματήσει η εκμετάλλευση της γεωργίας, η εξωτική βιομηχανία, η δική μας, ε, η διαφθορά της κυβέρνησης. Ε, εμείς φταίμε βρώμικα χέρια. Του κλέβουμε. Του κλέβουμε τι πλουτοπαραγωγικέ πηγέ. Είναι τόσο φτωχέ οι χώρε αυτέ Γι' αυτό το λόγο Εμεί τι πρόχουμε ακόμη περισσότερο στη φτώχεια. Να σταματήσουμε να τις καταλαιστεύουμε αυτές τις χώρες. Ε, επεκτατισμός, ε, τίποτα δεν κάναμε. Και όσα χρήματα και ρίξαμε εκεί πέρα. Να βοηθήσουμε την κυβέρνηση να σταχθεί στα πόδια τη, να σταματήσουμε να καταλαιστεύουμε τι χώρε αυτέ, να ξαναγίνουν φυσιολογικέ. Το λόγο έχει ο κύριος Πόλτσακ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να απευθύνω έκκληση υποστήριξη ε, για την Μπουρκίνα Φάσο. Η χώρα αυτή υποφέρει. Οι τσιχαντιστέ με τη βία του οδηγούν σε κατάρρευση το εσωτερικό σύστημα τη χώρας. Ε, δεν λειτουργεί πλέον τίποτα. Ε, η βία κατά των χριστιανών, κατά των παιδιών, των γυναικών είναι κάτι που πρέπει να το εμποδίσουμε. Θα πρέπει να στηρίξουμε τις εσωτερικές δονές της χώρας, ώστε οι ιδιοκτικές δυνάμεις να μπορέσουν να αναλάβουν δράση και όχι μόνο οι ένοπλοι ε, τρομοκράτες. και η ξηρασία ε, έχει οδηγήσει στη χώρα ε, σε αύξηση και ένταση των φαινομένων ε, φτώχειας. Πολλοί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι υποφέρουν. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε τη στρατηγική μας για ολόκληρη την περιοχή του Σαχέλ, όλες τις χώρες εκεί και να τις υποστηρίξουμε. Του το λόγο έχει εξ ονόμα της Επιτροπής ο κύριος Μπορέλ Φοντέλιες. Παρακαλώ. You have the floor. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, έχετε όλοι δίκιο. Τους τελευταίους μήνες έγιναν ε, μάρτυρες αυτές τις συνεχούς επιδείνωσης όσον αφορά την ασφάλεια στην Μπουρκίνα Φάσο. Και έχω διαβάσει ένα σωρό στοιχεία ακόμα περισσότερο από αυτά τα οποία εσείς είπατε. 700 είναι τα θύματα και 500 μόλις από το καλοκαίρι και έχουμε πάρα πολλές επιθέσεις διαφόρων ειδών κατά των διοικητικών αρχών, κατά των πολιτών, κατά χωριών και πόλεων. Και έτσι φτάνουμε σε 600, σε 700 χιλιάδες και περίπου εκτοπισμένους. Οπότε αυτή η κατάσταση σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε κρίση, οπότε ο κόσμος εκεί χρειάζεται βοήθεια, χρειάζονται κάποιες κοινωνικές ε, παροχές. Είναι πάνω από ένα εκατομμύριο εκείνοι οι οποίοι ε, χρειάζονται ήδη διατροφής. Και το καλοκαίρι είχαμε πάνω από 2.000 ε, σχολεία τα οποία έκλεισαν. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 300.000 ε, παιδιά τώρα στερούνται την μόρφωση και έχουμε περίπου 10.000 δάσκαλοι έχουν πληγεί, πολλοί έχουν σκοτωθεί φέτος έτσι αποδυναμώνεται η κυβέρνηση, θα έχουμε προεδρικές εκλογές σύντομα και θα πρέπει να υπόψη ότι άρχισαν ε, οι επικρίσεις ε, κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση που κάνει στο θέμα. Για εμάς είναι ένας ισχυρός εταίρος η χώρα και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες που αναδύθηκαν ε, πρόσφατα όσον αφορά την αξιολόγηση της κρίσης. Νομίζω ότι θα πρέπει η παρουσία μας εκεί να είναι πιο αποφασιστική στην περιοχή γενικότερα. Και 25% του πληθυσμού είναι οι χριστιανοί. Πολλέ φορέ αναφέρει τη χώρα ω παράδειγμα η μίμηση για ειρηνική συνύπαρξη. Όμω οι τρομοκρατέ εκεί θέλουν να υπονομεύσουν ε, αυτήν την ειρηνική συνύπαρξη, διότι υπάρχει μια ευρύτερη στρατηγική του όσον αφορά ε, τις προστριβές της ε, σύγκρουση και έτσι συνεχίζεται η εκτόπιση του πληθυσμού επιτίθεται σε κάποιες κοινότητες που τις θεωρούν εχθρικές αλλά επιτίθεται και σε μουσουλμάνους αυτοί που θεωρούνται πολύ μετριόφρονες, μετριοπαθείς από τους ε, τζιχαντιστές ε, έχουν επιτεθεί και σε τζαμιά το, τώρα το Σεπτέμβριο. Οπότε αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνουμε είναι κατεπηγόντως και αποφασιστικά να αναλάβουμε δράση όσοι έχουν προσυπογράψει ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα η χώρα αυτή θα πρέπει να βοηθεί από την διεθνή κοινότητα είναι υποχρέωσή της ούτω ώστε να δοθεί κάποια αξιοπρέπεια στον πληθυσμό της ε, χώρας και να εξασφαλιστεί η ελευθερία των θρησκευτικών πεπιθήσεων. Εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις και παρεμβαίνουμε εκεί που υπάρχει θέμα ε, ασφαλείας. Πρέπει να βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν την ριζοσπαστικοποίηση, να υπάρξει πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων, αλλά χρειάζονται χρηματοδοτήσεις και δώσαμε στις χώρες του Σαχέλ 10 εκατομμύρια για να υπάρξει και πάλι ειρηνική συνύπαρξη. Να βοηθήσουμε με άλλα 7 εκατομμύρια είπαμε την κοινωνία των πολιτών. Αυτά θα τα αναφέρω ενδεικτικά. Να τι κάνουμε σε αυτό το μέτωπο να υπάρξει κοινωνική συνοχή και θρησκευτική συνύπαρξη. Ε, έτσι θα εξασφαλιστεί η σταθερότητα στην χώρα. Σας βεβαιώ ότι θα συνεχίσουμε να βοηθούμε την χώρα να αντιμετωπίσει αυτή την κρίσιμη κατάσταση που αφορά γενικότερα την περιοχή του Σαχέλ και αφορά επίσης και την δική μας ασφαλεία και ειρηνικές προοπτικέ. Σας ευχαριστώ που φωτίσατε αυτό το θλιβερό πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Η συζήτηση έληξε. Ε, έλαβα 7 προτάσεις ψηφίσματος για την περάτωση αυτής της συζήτησης. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα. Η επόμενη συζήτηση στην ημερήσια διάταξη αφορά το Αφγανιστάν και συγκεκριμένα τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση αγοριών στην επαρχία Λογκάρ. Σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε να ζητήσετε το λόγο για το Catch the Eye και την μπλε κάρτα με δύο τρόπους. Με το συνήθι τρόπο, όσο και με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής, οι σχετικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στην είσοδο του ημικυκλίου. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Τσαρνέσκι. Ε, Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, ε, Κύριε είπατε εκπρόσωπε, χαίρομαι που πάνω από τις διαχωριστικές γραμμές των κομμάτων μιλούμε από καινού για αυτό το οδυνηρό ζήτημα, διότι η σεξουαλική κακοποίηση εις βάρος ανηλίκων είναι κάτι το αποτρόπαιο. Οπότε και πιστεύω ότι η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλες αυτές τις περιπτώσεις κακοποίησης στο Λογκάρ θα πρέπει να ακουστεί γιατί θα πρέπει να πιέσουμε την κυβέρνηση της χώρας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ανθρωπιστική οικονομική βοήθεια που δέχονται από την Ευρώπη. Άρα να τους πιέσουμε να κάνουν ό,τι μπορούν ούτως ώστε να σταματήσουν αυτές οι πρακτικές. Να περιοριστεί αυτή η κακοποίηση των ε, ανηλίκων. Είναι στίγμα ισόβιο αυτό το φαινόμενο. Αλληλεγγύη, να επιδείξουμε και χαίρομαι που υπάρχει διακομματικά κοινή θέση. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο κύριος Μπορέλ θα τοποθετηθεί διότι είναι ο πιο έμπειρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα αυτά. Το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Μαρκουάρτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω πάντα ένα πρόβλημα. Όταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάμε για το Αφγανιστάν, συζητάμε μόνο για τις σκοτεινές πλευρές. Το ξέρω ότι έχει σκοτεινές πλευρές το Αφγανιστάν, αλλά καμιά φορά καλό θα ήταν να συζητάμε και για τα ευχάριστα, για ευτυχισμένες οικογένειες, για το μας στην Καμπούλ, για το ωραίο φαγητό. Το ξέρω ότι δεν είναι αυτό το θέμα μας, αλλά είναι θλιβερό γιατί ακούμε μόνο τα σκούρα, τα μαύρα. Το 16 και το 17 ήμουν ως δημοσιογράφος στο Αφγανιστάν και είδα και τα σκοτεινά, αλλά γνώρισα και καταπληκτικούς ανθρώπους, πολλούς, που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Όπως ο Μοχάμετ Μούσα Μαχμούντι και άλλοι οι οποίοι ακούραστα αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αξίζει να τους ευχαριστούμε. Και... κρίμα που οι αγωνιστές και ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προστατεύονται λιγότερο από κάποιου αξιωματούχους... που εγκληματούν κατά παιδιών. Τα κακοποιούν σε, σεξουαλικά. Και, ε, καλό είναι λοιπόν που λέμε το θέμα και υπήρξαν και κάποιες συλλήψεις ε, ε, κάποιων αξιωματούχων που πρόκειται να συναντηθούν με ένα ε, πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό είναι να εξετάσουμε αυτές τις περιπτώσεις ανεξάρτητα, αλλά να μην χάσουμε την εικόνα, να δούμε πραγματικά τι γίνεται στο Αφγανιστάν, να μην παραμένουν αυτά τα εγκλήματα ατιμόρυτα, αλλά να προστατεύονται και οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και όποιο θέλει να πάρει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθάει τους αγωνιστές και ε, ε, θα πρέπει να φροντίζει να διώκονται οι εγκληματίε κατά των παιδιών. Στο ψήφισμα αναφέρουμε διάφορα θέματα και χαίρομαι και είμαι πολύ ευγνώμων που καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα ευρύ ψήφισμα για να στείλουμε και ισχυρά μηνύματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Πύρη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή είναι μια βάναυση εικόνα που όλους ε, μας σόκαρε. Ε, αξιωματούχοι του Αφγανιστάν παίρνουν παιδιά από ε, τι οικογένειέ του, τα δίνουν γυναίκες, γυναίκε, τα μάθανε να χορεύουν και μετά τα κακοποιούν σεξουαλικά. Το είναι το μπακαμπάζι. Αλλά δεν πρέπει να μένουμε στι λέξει. Μιλάμε και σεξουαλική σκλαβιά. Και πρέπει να τιμωρείται. Είναι επιλήψιμο και, και κολάσιμο. Ε, τουλάχιστον 1.300 παιδιά, αγόρια στην περιοχή Λογκάρ και χιλιάδες παραπάνω σίγουρα που δεν γνωρίζουμε έχουν καταγραφεί ότι ειδοποιήθηκαν σεξουαλικά στα σχολεία τους από τις αρχές. Κάποια θανατώθηκαν, πέντε από τις οικογένειες γιατί έφεραν ντροπή στις κοινότητές τους. Οι αφγανικές αρχές πρέπει αμέσως να αναστείλουν, να συλλάβουν όλες, όλους τους δράστες της πρακτικής αυτής του Μπακαμπάζη και να κάνουν ανακρίσεις και έρευνες για όλες τις υποθέσεις, ώστε οι αυτουργοί, οι υπεύθυνοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Το λόγο έχει η κυρία Ματίας για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υποστηρίζουμε αυτό το ψήφισμα πλήρω. Οι περιπτώσει σεξουαλική κακοποίηση είναι μια από τι πιο απαράδεκτε καταστάσει. Θα πρέπει στο Αφγανιστάν να παραδεχτούμε ότι δεν ήταν ποτέ τα πράγματα πολύ καλά, αλλά εδώ υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι 36 νέοι είναι ε, μια από τις περιπτώσεις που ε, μεταξύ του 2015 και 2018 μας δείχνει ότι εκατοντάδες παιδιά κακοποιήθηκαν στο Αφγανιστάν. Το φαινόμενο όμως έχει μεγαλύτερες διαστάσεις και θα πρέπει να καλέσουμε τους συναδέλφους να στηρίξουν τις τροπολογίες που βάλουμε στο ψήφισμα. Υποστηρίζουμε πλήρως το ψήφισμα αλλά προσθέτουμε στο πλαίσιο της ε, δράσης μας ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτό που επιβεβαίωσε ο ειδικό επιτετραμένο τον είπα ε, στην περιοχή. Ότι οι δυνάμει των ΗΠΑ δεν παρενέβησαν σε αυτέ τι περιπτώσει κακοποίηση ε, και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρουμε ότι οι Αμερικανικέ δυνάμει ε, ε, ουσιαστικά εθελοτυφλούσαν στι περιπτώσει κατάχρηση εξουσία των Αφγανικών αρχών. Υπήρξαν παραβιάσει τι οποίε οργάνωσαν παραστατικέ ομάδε και που υποστήριζαν οι ΗΠΑ. Τώρα που όλοι τα γνωρίζουμε αυτά, που έχουν γνωστοποιηθεί, πρέπει να προσθεθεί στο ψήφισμα η ανάγκη να γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα ώστε να μην παραμείνουν σε ατιμορρησία όσοι τα διέπραξαν. Και στο ψήφισμα αυτό καλούμε τα κράτη-μέλη να ε, φροντίσουν να μην επιστρέψουν ε, και απελαθούν νέοι Αφγανοί που όταν επιστρέψουν στη χώρα αντιμετωπίζουν αυτή τη φρικτή πραγματικότητα που δείχνει το ψήφισμα. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Οστρεβίτσιους. Πρόεδρε, κύριε Πατεκπρόσωπε, αγαπητοί συνάδελφοι, τα εγκλήματα κατά των παιδιών είναι τα χειρότερα εγκλήματα. Καταστρέφουν και τους αφαιρούν την παιδική τους ηλικία σε αυτά τα παιδιά τα μικρά από το Αφγανιστάν. Και επιπλέον επηρεάζει και τη ζωή τους και το μέλλον τους αυτό. Το μέλλον τους είναι το μέλλον του Αφγανιστάν που εργαζόμαστε σκληρά για να δημιουργήσουμε. Τις τελευταίες μέρες είδαμε ότι δεσμεύτηκε ο πρόεδρος Γκάνη να διερευνηθούν αυτά τα φρικτά που γίνονται στα σχολεία στην επαρχία Λογκάρ. Χαιρόμαστε για την αντίδραση αυτή και προσβλέπουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όλοι οι δράστες θα πρέπει να παραπευθούν στη δικαιοσύνη και τα σχολεία να ξαναγίνουν ένα ασφαλές μέρος για τα παιδιά. Ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι η ενοικοδόμηση του Αφγανιστάν για να υπάρχει ασφαλές ε, μέλλον για τη νέα γενιά της χώρας. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την προσπάθεια εξολόθρευσης ε, της πρακτικής Μπαχαμπασί και να προστατεύουμε τα δικαιώματα των παιδιών στο Αφγανιστάν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για δύο λεπτά η κυρία Ζόβκο. Κύριε Πρόεδρε, πριν από μόλις λίγες εβδομάδες είχαμε την 30η επέτειο για την Συνδίκη των δικαιωμάτων του παιδιού και με την σημερινή συζήτηση ολοκληρώνουμε ε, το, το πλέγμα αυτό προστασία για τα παιδιά σε όλο τον κόσμο. Προβληματιζόμαστε βαθιά όσον αφορά αυτού του ε, ισχυρισμού, τι καταγγελίε για κακοποίηση σε πολλά μέρη του Αφγανιστάν. Προστασία του παιδιού θα πρέπει να είναι μέλημα κάθε κοινωνία, ιδίω όταν υπάρχουν ένοπλε συγκρούσει. Επίση, ε, καταδικάζουμε το ότι έχουν φυλακιστεί διάφοροι ακτιβιστές ανθρώπινων δικαιωμάτων που καταγγέλουν τέτοια συμβάντα. Οι αρχές της χώρας θα πρέπει να εξασφαλίσουν σε κάθε περίπτωση ότι αυτοί οι ακτιβιστές των δικαιωμάτων θα μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους. Οπότε έρχομαι τώρα να ε, πω στο ότι ο Ευρωπαίος Αγγελέας θα πρέπει να διερευνήσει αυτούς τους ισχυρισμού αλλά και αυτές τις αυθαίρετες φυλακίσεις των ακτιβιστών. Η αντιπροσωπεία μας, ε, οι χώρες μας, η διπλωματία μας θα πρέπει να παρακολουθήσει τις εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση και να υλοποιήσει τις κατευθυντήριες όσον αφορά την προστασία των ε, ανηλίκων σε καιρό πολέμου. Επίσης, πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να ελέγξει, να παρακολουθήσει, να υποπτεύσει τι γίνεται με την οικονομική μας ενίσχυση προς τη χώρα. Και έτσι θα εξασφαλίσουμε ότι αυτή η χρηματοδότηση θα βοηθήσει στο να υπάρχει περιβάλλον προστασίας για τα παιδιά και για τους ακτιβιστέ. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Προχωρούμε στον κύκλο των ομιλητών εκ μέρου των πολιτικών ομάδων για την ομάδα της των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών. Το λόγο έχει η κυρία Σάντος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κατάσταση που συζητούμε εδώ, γι' αυτό το ε, έθιμο, το έθιμο που είναι φρικτό του Μπαχαμπαζή στο Αφγανιστάν, ουσιαστικά προκαλεί έντονη απέχθεια. Είναι μια παράδοση που υπάρχει από πάντα στη χώρα, αλλά πραγματικά αποτελεί παραβίαση των παιδικών δικαιωμάτων και των βασικότερων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας και υποσχέσεις του Αφγανιστάν για την εκρίζωση αυτού του φαινομένου είναι αναπαρκή. Ε, εδώ θα πρέπει να, να δούμε τις μαρτυρίες αγοριών που έχουν κοκοποιηθεί και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν δεχθεί επίθεση και αυθερέτως έχουν κρατηθεί φυλακιστεί. Πρέπει λοιπόν να απαιτήσουμε απελευθέρωση όλων όσοι εργάζονται για τα δικαιώματα των παιδιών και θα πρέπει να υπάρξει πλήρης εκρίζωση αυτής της πρακτικής κακοποίησης πρέπει να προβλέψουμε ένα τέλος για το καθεστώς ατιμορρησίας και να έχουν πρόσβαση αυτά τα παιδιά στο σύστημα δικαιοσύνης και να μην υπάρξει απέλασή τους όταν φτάνουν ως τις χώρες μας. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι διαδικασίες καθυστερούν ε, και αυτό επειδή υπάρχει κινητοποίηση στην κοινωνία των πολιτών στο Αφγανιστάν, θρησκευτικών ηγετών, ε, πολιτών. Όλοι χρειάζονται για να καταπολεμήσουμε αυτή τη μάστιγα και χρειάζεται και μια νομοθετική μεταρρύθμιση, αλλά σαφώ και παρέμβαση μέσω του εκπαιδευτικού συστήματο, ώστε να προστατευτούν οι μελλοντικέ γενιέ. Σα ευχαριστώ. Για την ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας, το λόγο έχει η κυρία Άντερσον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η κακοποίηση των παιδιών στο Αφγανιστάν είναι αποτρόπαια. Η σεξουαλική κακοποίηση κάθε παιδιού είναι αποτρόπαια. Δυστυχώς, αυτό το είδος κακοποίησης ε, συνηθίζεται στις Ισλαμικές χώρες. Και άλλωστε ε, είναι έκφραση της κυρίαρχης κουλτούρας εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δείχνει τώρα μια ξυπασιά και το δάχτυλο στα στρεβλά άλλων κρατών. Πάλι κηρύγματα κυριακάτικα και λόγια, κούφια. Ε, για να αποδείξουμε την ηθική μας ανατερότητα. Αλλά τι θα αλλάξετε στην πραγματικότητα που ζουν αυτά τα παιδιά. Και μόνο ε, αν ε, το αναφέρει, αν αναφέρει κανείς ότι φταίει το Ισλάμ, σε λένε ρατσιστή εδώ. Δεν μπορούμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μην καμώνεστε τώρα ότι σας νοιάζει και η μοίρα των παιδιών αυτών. Ε, αυτή η ηθική αναθεω, ε, ανωτερότητα είναι κάτι το οποίο περιφέρεται ε, και είναι τρομερή υποκρισία. Για την ομάδα Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, το λόγο έχει η κυρία Ντέλη για δύο λεπτά. Thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω το ψήφισμα αυτό από τη σκοπιά ε, της ε, επανάληψης της συζήτησης για την αποτρόπαια πρακτική του Μπαχαμπάζε, τη συστημική, ε, την συστηματική μάλλον σκλαβιά γοριών στο Αφγανιστάν και τη σεξουαλική τους κακοποίηση. Είναι θλιβερό αυτό. Το θλιβερότερο όμως στην όλη συζήτηση είναι ότι δεν πρόκειται περί αποκάλυψη, δε, ε, αποκάλυψης, δεν είναι κάτι καινούριο. Το γνωρίζαμε από πάντα και στην πραγματικότητα γνωρίζουμε ότι κάθε απόπειρα να αποκαλυφθεί η κατάσταση και να αντιμετωπιστεί έχουν ε, παρακολουθεί. Ακόμα και Αμερικανοί στρατιώτες προσπάθησαν να εμποδίσουν την πρακτική. Και αυτοί οι ίδιοι δέχτηκαν ε, πειθαρχικές ε, προειδοποίησεις. Άλλωστε, πολλέ φορέ στρατιώτε διέπραταν αυτέ τι πρακτικέ με παρουσία και ανοχή των Αμερικανών. Η αμερικανική παρουσία στι ΗΠΑ, λοιπόν, υποτίθεται ότι ήθελε να φέρει ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών και δικαιώματα στην εκπαίδευση. Όμω η πρακτική αυτή ε, μπορούσε να διαπράσετε με την ανοχή τους και δεν έκαναν τίποτα. Θα πρέπει όλες οι υποθέσεις να ερευνηθούν και όλα τα θύματα να έχουν την ανάλογη υποστήριξη και προστασία. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει να αντλήσουμε και τα κατάλληλα διδάγματα. Είναι πραγματικά ε, θλιβερό το μήνυμα ότι εδώ ε, καταδικάζουμε τη σωματική φυλάκιση και κακοποίηση των ε, παιδιών, ενώ όλη η χώρα έχει κακοποιηθεί, σκλαβωθεί και φυλακιστεί από ξένε δυνάμει. Το Αφγανιστάν είναι από τι πιο βίαιε χώρε στον κόσμο. Και όμω εμεί στέλνουμε εκατοντάδε νέου πίσω κάθε χρόνο. Το κοινοβούλιο λέει ότι είναι ανασφαλή χώρα για να την επισκεφθούμε. Όμω εμεί επιστρέφουμε τα παιδιά τη χώρα πίσω κάθε χρόνο. Κακώ θα πρέπει να υπερασπιστούμε το δικαίωμά του να ζουν αξιοπρεπώ στη χώρα του, αντί να παρεμβαίνουμε με βιαιότητα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ειρήνευση στη χώρα, ναι μεν, αλλά θα πρέπει να προσπιστούμε κυρίω του ακτιβιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλου του πολίτε εκεί που δρούν και όχι τι επίσημε αρχέ. Επόμενο εγγεγραμμένο ομιλητή είναι ο κύριο Καστάλντο, τον οποίο δεν βλέπω παρόντα στην αίθουσα. Επομένω, το λόγο έχει ο κύριο Μπιεντρών για ένα λεπτό. Φανταστείτε ένα νεαρό αγόρι, 13, πάει σχολείο για να μορφωθεί, όπως το αξίζει. Φανταστείτε ο δάσκαλός του, που τον εμπιστεύεται αυτό το παιδί, το οδηγεί σε μια σκοτεινή αίθουσα και το βιάζει. Το αγόρι είναι θεραλέο. Καταγγέλει αυτό που συνέβη. Αλλά αν πάει σε ένα αστυνομικό τμήμα, ξαναβιάζεται. Η οικογένεια του παιδιού αισθάνεται τέτοια ντροπή που τον πετάνε έξω. Αλλά τουλάχιστον δεν τον σκοτώνουν. Αυτή η περίπτωση δεν είναι μεμονωμένη. Ε, είναι εκατοντάδε οι υποθέσει αυτέ που έχουν επαληθευτεί στην αυγανική περιοχή του Λογκάρο, όπου οι δάσκαλοι και οι τοπικοί αστυνομικοί έχουν εμπλακεί σε ένα δίκτυο παιδεραστία. Και τώρα φανταστείτε να μην κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Εντσίρ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή και το ψήφισμα αυτό ε, πραγματικά ε, είναι ό,τι χειρότερο μπορούσαμε να φανταστούμε. Ένα πηγάδι χωρίς ε, πάτο. Εδώ λοιπόν δεν φαίνεται να βρίσκουμε να μπορούμε να περιοριστούμε μόνο σε ένα ψήφισμα. Πρέπει να θέσουμε το θέμα σε οποιοδήποτε πολιτικό επίπεδο. Σεξουαλική κακοποίηση, δολοφονία, εμπορία αγοριών, νέων παιδιών είναι αρρωστημένο, είναι απαράδεκτο. Ε, η κατάσταση των αγοριών στην αφγανική περιοχή του Λογκάρ είναι σκανδαλώδη. Θέλω λοιπόν να εκφράσω την πλήρη αλληλεγγύη μου προ τα θύματα. Πρέπει να πάψει η κουλτούρα, η κουλτούρα της ε, σιωπής και της ντροπή για την πρακτική αυτή μπαχαμπάζη. Πρέπει να πάψουν αυτά και πρέπει όλοι οι υπεύθυνοι να συρθούν στη δικαιοσύνη. Πρέπει να αναλάβουν τι ευθύνε του. Το δικαστικό σύστημα πρέπει επιτέλου να λειτουργήσει και οι νέοι πρέπει να έχουν τη στήριξη και τη βοήθεια που του αξίζει. Έχουν δικαίωμα σε αυτό. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να είναι παιδιά και να μεγαλώσουν ε, κανονικά, ήρεμα και χωρί τέτοιε βάναυσε ε, ε καταστάσει. Ευχαριστώ ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των εγγεγραμμένων ομιλητών. Προχωρούμε στη διαδικασία του Catch the Eye. Έχω δεχτεί τρία αιτήματα. Γίνονται και τα τρία αποδεκτά. Το λόγο έχει ο κύριος Πόσπισιλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι φρικτά αυτά τα οποία γίνονται στο Λογάρ δεν περιγράφονται αυτά που γίνεται τον των ανηλίκων. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Κύριε, είπατε εκπρόσωπε, πρέπει να ασκηθεί η οικονομική πίεση και όχι μόνο προς την κυβέρνηση. Να δουν το ζήτημα σοβαρά, να το αντιμετωπίσουν, όχι άλλες υποσχέσεις. Και πρόσφατα τα ξανασυζητήσαμε. Η εξωτερική μας πολιτική θα πρέπει να το δει σοβαρά. Σας ζητώ να απαιτήσετε από την χώρα να λάβει μέτρα να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της σεξουαλικής βίας, να γίνει διερεύνηση και να σύρουν ενώπιον της δικαιοσύνης τους ενόχους, να μπει ένα τέρμα σε αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει να μην επανελθούν αυτά τα φαινόμενα. Και φοβάμαι ότι αλλιώς τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι. Ε, ε, βλέπουμε από τις τελευταίες εκθέσεις του ΟΗΕ ότι χιλιάδες παιδιών ε, δολοφονούνται ή ακροτηριάζονται. Υπάρχει και σωματική βία κατά των ανηλίκων στο Αφγανιστάν και δυστυχώς παρόλα τα μέτρα που έχουν γίνει με τη νέα νομοθεσία και το νέο ε, ποινικό κώδικα το 2016 για τα δικαιώματα των παιδιών. Όλα αυτά ήταν μάταια. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπερψηφίσουμε ε, σήμερα το συγκεκριμένο ψήφισμα. Υπάρχει μια τροπολογία όπου καταδικάζεται ρητά και απερίφραστα η πρακτική των ξένων στρατευμάτων. Δεν έχει γίνει τίποτα εκεί κακοποίηση παιδιών έχουμε και στα δικά μας κράτη-μέλη. Έχουμε ανηλίκους που κακοποιούνται και στη δική μου χώρα. Πρόσφατα είχαμε τέτοια φαινόμενα. Αλλά τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Θα πρέπει να τα προσέχουμε, να τα φροντίζουμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Ε, ολοκληρώθηκε. Ε, μάλλον, ε, σας καλημερίζω και σας και τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών που μας παρακολουθούν. Ε, δίνω το λόγο στον κύριο Μπάλλα, από, μάλλον στον κύριο Γόλα από την ΚΟΕ. Um, uh, Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αυτό το φαινόμενο της κακοποίησης παιδιών θα πρέπει να είναι από τα φρικτότερα που μπορεί κανεί να βάλει στο μυαλό του. Εγώ προέρχομαι από την Ιρλανδία και έχουμε και εκεί σεξουαλική κακοποίηση νέων από κάποιου ε, ιερεί καθολικού και αυτό είναι καταστροφικό στη χώρα μας ήταν γνωστό ότι αυτό συνέβαινε αλλά ήταν τα στόματα φημωμένα, κλειστά και φοβάμαι ότι το κατεστημένο και η κυβέρνηση του Αφγανιστάν επίσης αποκλείεται να μην γνωρίζουν. Άρα θα πρέπει εμείς να βοηθήσουμε να στηρίξει τα πόδια της η χώρα αφού την κατέστρεψαν οι Ρώσοι και μετά οι Αμερικανοί. Αλλά αν θέλουμε ο ρόλος μας να είναι θετικός θα πρέπει να είμαστε αυστηροί. Θα πούμε έξω τα δόντια στην κυβέρνηση. Δεν είναι δυνατόν τέτοια πράγματα να είναι αποδεκτά. Με την σιωπή δεν έρχεται η αλλαγή. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ειδικό μας βάρος ούτως ώστε να ακουστεί εκεί η φωνή μας ότι αυτά τα πράγματα παρά είναι δυσάρεστα, καταστροφικά. Κύριε Μπουρέλη, έχετε το λόγο. Ε, αξιότιμα μέλη, φυσικά στις ε, ανεπτυγμένες και ε, πλούσιες κοινωνίες μας υπάρχουν φαινόμενα κακοποίησης παιδιών. Αλίμονο. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και τον πόλεμο στο Αφγανιστάν και για ποιο λόγο έχουμε πάει και εμείς οι Δυτικοί για μια εικοσαετία και πλέον. Ποια ήταν τα αίτια, τα αποτελέσματα, όλα αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε όποτε θέλετε. Αλλά αυτό που σήμερα μας απασχολεί είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση. η οποία είναι η κορυφή του παγόβουνου. Τα δεδομένα που έχουμε και τα στοιχεία ε, για κακοποίησης παιδιών στο Αφγανιστάν δυστυχώς είναι απείρως περισσότερα και ούτε ε, υπάρχει καμία σύγκριση με τις δικές μας κοινωνίες. Δείχνουν λοιπόν τα στοιχεία που έχουμε ότι η περίπτωση Λογκάρ είναι ακριβώς η κορυφή του παγόβουνου, η ορατή. Από το 2015 μέχρι το 2018 η Task Force των Ηνωμένων Εθνών εντόπισε 40.000, 40.000 σοβαρές παραβιάσεις και κακοποίησεις κατά των παιδιών σε όλη τη χώρα. Πολλές από αυτές μας ανησυχούν βαθιά και αφορούν 80% των αμάχων θυμάτων των παιδιών. Παρόλη την παρακολούθηση που είναι δύσκολη και την επαλήθευση, 274 παιδιά έχουν κακοποιηθεί σοβαρά απάγονται, κακοποιούνται, βιάζονται 800 και τα λοιπά σε νοσοκομεία και σχολεία είναι γνωστά τα προβλήματα αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συγκριθούν με τόσα συμβαίνουν εδώ στο Αφγανιστάν το 2017 θέλησαν να αναθεωρήσουν τον ποινικό κώδικα ο οποίος ετέθη σε ισχύ το 2018 και ρητά ποινικοποιεί αυτή την πρακτική τη λεγόμενη μπαχαμπάζη. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο καμιά φορά να αλλάξουν οι συνθήκες, η επιρροή κάποιων ισχυρών και η τιμωρησία είναι ευρύτατα διαδεδομένη. Τα δε θύματα στιγματίζονται και αποκλείονται από την κοινωνία. Θα πρέπει να αγωνιστούμε γιατί η προστασία των παιδιών κανονικά έπρεπε να εγκριθεί και από προεδρικό διάταγμα. Και αργότερα η κάτω βουλή του Κοινοβουλίου αρνήθηκε να το εγκρίνει γιατί λέει δεν υπήρχε απαρτία για να εγκριθεί ένα άρθρο. Και το Δεκέμβρη του 2019 στις 11 του μηνός, της προάλλης δηλαδή, ακόμα συζητούσαν αυτό το θέμα για την προστασία των παιδιών και τον νόμο για τα δικαιώματα των παιδιών. Τέσσερις φορές ο νόμος αυτός στην τελευταία τετραετία περίφθη από το Κοινοβούλιο. Δείχνει πόσο ισχυρές είναι οι αντιστάσεις για να αλλάξει η νομοθεσία και βασικά οι συνήθειες και τα έθιμα και τα ήθη σε μια κοινωνία που δυστυχώς ε, εμφανίζει τέτοιες συμπεριφορές. Αυτές θα πρέπει να καταπολεμηθούν και πρέπει εμείς να βοηθήσουμε στην καταπολέμησή τους να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τα δικαιώματα των παιδιών στο Αφγανιστάν. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και θα εξακολουθήσουμε να το πράττουμε αυτό, γνωρίζοντας ότι τελικά για να αλλάξει μια κοινωνία χρειάζονται πολύ μεγάλες προσπάθειες. Είναι μακράς πνοής αυτή η προσπάθεια. Δεν αρκεί να περάσει μια νομοθεσία και να δημοσιευθεί σε μια επίσημη εφημερίδα. Πρόσφατα διοργανώσαμε δημόσια διαβούλευση με τίτλο «Τα παιδιά του Αφγανιστάν» αξίζουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό γέννησε μεγάλο ενδιαφέρον από εξαρματούχους και το γενικό κοινό και έχουμε και ένα ετήσιο διάλογο για τα δικαιώματα με την αφγανική κυβέρνηση και εκεί συστηματικά εντάσσουμε ένα κεφάλαιο για την ειδική κατάσταση των παιδιών όπου τέτοια πράγματα μας απασχολούν η βία κατά των παιδιών, η κακοποίηση, το μπαχαμπάζι και η αναγκαστική γάμη. Βεβαίω υπάρχουν ε, περιπτώσεις καταχρήσεων και στις ένοπλες δυνάμεις. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση συστηματικά θέτει υπόψη των συνομιλητών της αυτό το θέμα για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι ε, προσλήψεις, στρατολογούνται οι ε, στρατιωτικοί και για τη συμπεριφορά των αστυνομικών κατά του αμάχου γενικού πληθυσμού. Υπάρχει και ε, παροχή συμβουλών εκεί, ακριβώς και προς όφελος των ε, ανελίκων και των νέων. Όπως βλέπετε είναι τεράστιο το πρόβλημα. Εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις ε, αφγανικές αρχές και την κοινωνία να το καταπολεμούν. είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναφέρει αυτά τα φαινόμενα για να μπορέσουμε να τα καταπολεμήσουμε. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και σας ενημερώνω ότι Έχω λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος, τις οποίες θα ψηφίσουμε στη συνέχεια. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι ο ρωσικός νόμος περί ξένων πρακτόρων. Έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο και γι' αυτό σας παρακαλώ να μην ε, υπερβείτε το ένα λεπτό. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Φωτίγκα. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε και κύριε είπατε εκπρόσωπε, η Σοβιετική Ένωση ήταν ιδιαίτερα κατασταλτική, κατεπιεστική, βάναυση σε σχέση με την εξάρτητη δημοσιογραφία. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν, εξοντώθηκαν και βλέπουμε τώρα στη Ρωσική Ομοσπονδία ότι γίνονται διάφορα από το κράτος τα οποία μας θυμίζουν δυστυχώς το παρελθόν. Θυμόμαστε ακόμα την ε, πολιτικόσκαγια άλλους θωραλέους ε, δημοσιογράφους οι οποίοι ήθελαν να υπάρξει αντικειμενική ενημέρωση για την ε, Ρωσία. Δυστυχώς αυτή η νομοθεσία για τους ξένους πράκτορες του Βλάντιμιρ Πούτιν της ε, ε, Δευτέρας Δεκεμβρίου αποσκοπεί στο να εκφοβήσει τους ε, bloggers και τους δημοσιογράφους. Και θέλουμε αυτό το ψήφισμα να ζητήσουμε την κατάργηση αυτού του νόμου. Φων Κράμον τον Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Για άλλη μια φορά ο Πούτιν θέλει με αυτή την νομοθεσία για ξένους πράκτορες να ε, ελέγξει ακόμα περισσότερο την κοινωνία του. Ο χώρος για ελευθερία της έκφρασης, μίντια κτλ. συρρυκνώνεται συνεχώς. Βήμα-βήμα φερεί το Κρεμλίνο κάθε ελευθερία από τους πολίτες. Δεν ισχύει αυτό μόνο στη Ρωσία είναι το καλύτερο εξαγωγικό προϊόν αυτό, Πούτιν ως ε, πρότυπο για αυταρχικούς ηγέτες. Δεν φυλακίζουν πάντα την αντιπολίτευση, αλλά έχουν καταλάβει ότι αρκούν τα διοικητικά μέτρα ή ακόμα και οι απειλές ε, έχουν ε, λεπτύνει, βελτιώσει τις μεθόδους τους για να ε, εκφοβίζουν και να φημώνουν τελικά και τις ΜΚΟ. Αυτό είναι καθημερινή πρακτική. Συγκρατίες συγκοφάντησης κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη Ρουμανία, Τσεχία και Μάλτα, όχι μόνο. Ο Βίκτορ Ορμπάν είναι ο πιο καλός ο μαθητής του Πούτιν στην ε, Ουγγαρία οι ΜΚΟ πρέπει να καταγράφονται και μάλιστα να λένε όταν παίρνουν χρήματα από το εξωτερικό να χαρακτηρίζονται ως οργανώσεις χρηματοδοτούμενες έξωθεν. Θα πρέπει αυτό να σταματήσει, να κόψουμε αυτές τις πρακτικές. Ε, Πίτσουλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου για την εξαιρετική συνεργασία και τι επικοδομητικέ διαπραγματεύσει. Είχαμε ένα πολύ καλό κοινό που βασίζεται στο όλο πρόβλημα και επικεντρώνεται στο όλο πρόβλημα των ξένων πρακτόρων του σχετικού νόμου. Είναι σαφέ το μήνυμα που στέλνουμε. Ο νόμο εγκρίθηκε το 2012, αλλά τον περασμένο μήνα πέρασαν καινούργιε τροπολογίε στον νόμο και τώρα θα αφορά ο νόμο όλου όσοι δημοσιεύουν περιεχόμενο ή ε, το ε, διανέμουν, ε, το διαδίδουν και δέχονται κονδύλια εκτός Ρωσικής Ομοσπονδίας. Εδώ περιορίζεται κι άλλο η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η δημοσιογράφη, η ελευθερία λόγου και έκφρασης και βεβαίως ό,τι περί μέσων μαζικής ενημέρωσης έχει να κάνει με το ρωσικό σύνταγμα. Θα πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα και η Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να γίνονται σεβαστή και από τη Ρωσία. Η Ρωσία πρέπει να ε, σεβαστεί τι αρχέ τη οποία έχει προσυπογράψει. Θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία. Θα πρέπει η Ρωσία να συμμετέχει σε μια σφαιρική στρατηγική για την τήρηση τη ε, παγκόσμια τάξη. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο συνάδελφο Κουκ. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει τίποτε σημαντικότερο για την δημοκρατία όπω η ελευθερία του λόγου και τίποτε σημαντικότερο από την ασφάλεια όπω η δημοκρατία στην Ευρώπη και γύρω από την Ευρώπη. Ο μεγαλύτερο από του γείτονέ μα όμω έχει ε, κάνει κι άλλο ένα βήμα που μα ανησυχεί. Η Ρωσία περιορίζει του συντάκτε ιστολογίων, του δημοσιογράφου και του ε, κατηγοριοποιεί ω ξένου πράκτορε. Απειλεί να του τιμωρήσει. Ε, αφορά την πλειοψηφία των μέσων μαζική ενημέρωση αυτό και όσοι δεν ε, συμφωνούν με την κυβέρνηση ε, θα απειλούνται με φυλάκιση. Με Η καταστολή Θέλουμε φιλικέ σχέσει με τη Ρωσία, όχι εχθρικέ. Όμω το ρωσικό καθεστώ δεν μπορεί παρά να επικριθεί. Και με τις ε, συχνές αλλαγές ε, της δημοκρατίας ε, στην κορυφή τη εξουσία, καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντικότερο, το σημαντικότερο η ελευθερία του λόγου. Δεν θέλουμε να υπάρχει αυτή η απειλή ούτε σε εμά ούτε στου γειτονέ μα. Και θα πρέπει η ανεξέλεγκτη αμοιβαία καχυποψία να πάψει. Να υπάρξει περισσότερη ελευθερία του λόγου και όχι λιγότερη στη Ρωσία. Ευχαριστούμε. Και τελευταίος από τους συντάκτες ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πραγματικά και πάλι δυστυχώ πρέπει να ασχοληθούμε με μια τροπολογία του νόμου στην Ρωσία. Δεν έχει, έχει να κάνει μάλλον με, με κυβερνητικέ οργανώσει που λαμβάνουν χρηματοδότηση εκτό Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό αφορά και του συντάκτε ιστολογίων, του blogger και ε, του δημοσιογράφου. Και βεβαίω είναι χτύπημα για την ελευθεροτυπία. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαφθορά. Ε, και πολύ εύκολα κατηγοροποιούνται οι δημοσιογράφοι ω ξένοι πράκτορε. Πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Το αξίζουν οι Ρώσοι πολίτε. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα πραγματικά συμφέροντα των πολιτών απέναντι σε μια μικρή πολιτική και οικονομική ελίτ και την κορυφή της πολιτικής εξουσίας της χώρας. Υπάρχει βεβαίως εθνικισμός στη χώρα, αλλά δεν υπήρξε καμία δυναστεία ε, στο παρελθόν της ιστορίας της Ρωσίας που μπορούσε να διοργανώσει έτσι την εξουσία, ώστε να υπάρχει μια πρόσωψη που θα τα επιτρέπει όλα σε αυτή την ελίτ. Εδώ λοιπόν πρέπει από αλληλεγγύη να εκφραστούμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρξει και χειροπιαστή υλοποίηση θα πρέπει να απαιτήσουμε την αναστολή του νόμου αυτού. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Κουμπίλιος. Πρώτα πρώτα θα πρέπει να απαντηθεί το εξής απλό ερώτημα. Τι ορίζει αυτός ο οριστικός νόμος ξένους πράκτορες. Σημαίνει ότι οι αρχές φοβούνται το λαό και γι' αυτό και θέλω να πω το εξή, μια έκκληση στον κύριο Πούτιν. Μην φοβάστε τον ε, Ρώσο απλό πολίτη. Τους φοβούνται και αρχίζουν να τους διώκουν. Ε, για αυτό και καθόνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, για αυτό και θα πρέπει να ασκήσουμε κάθε δύναμη επιρροής. Και ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως Συμβούλιο της Ευρώπης μια που τώρα ε, ανέκτησε εκεί την έδρα της η Ρωσία. Συμβούλιο, Κομισιόν, εμείς, οι κυβερνήσεις μας, στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Όλους, όλους να τους πείσουμε να ε, ταχθούν υπέρ των δικαιωμάτων των ε, Ρώσων κατά αυτών των αρχών που φοβούνται το λαό τους. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος και δίνει το λόγο στον κύριο Γκλούξμαν για τους Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε η Επιτροπή για την πρόληψη των βασανιστήριων είναι ξένοι πράκτορες. Η ομάδα Maximum για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, ξένος πράκτορ. Η ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μεμόρια, ξένο ξένος πράκτορ. Οι ε, οικολόγοι της Μπελώμα, ξένοι πράκτορες. Και τώρα και οι bloggers, δημοσιογράφοι, άτομα μεμονωμένα, διανοούμενοι, απλοί πολίτε, όλοι ξένοι πράκτορε. Αυτό το μοντέλο κοινωνία προτείνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ε, και αυτό εμπνέει όλα τα αυταρχικά καθεστώτα. Ας μην γελιόμαστε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι απλώς διπλωματικό το θέμα. Είναι η σύγκρουση δύο θεωρήσεων του κόσμου. Δύο κόσμο θεωριών. Και θα πρέπει, συνάδελφοι, να είμαστε συνεπείς ε, στην υπεράσπιση της δημοκρατίας όσο συνεπής είναι ο Πούτιν στις επανειλημμένες του επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και στη Ρωσία και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Οστρεβίσιους, παρακαλώ. Madam Chair, Representative for a long time... Επί πολύ χρόνο έχουν στριμώξει τα ανεξάρτητα μέσα οι ρωσικές αρχές. Πάρα πολύ λίγοι είναι πια οι αξιόπιστοι, δημοσιογράφοι αξιόπιστες πηγές. Τώρα φύγονται συγκεκριμένα πρόσωπα, ε, όλοι αυτοί που είναι αντιπολίτευση και εκτιβιστές που διαφωνούν με το όραμα του Κρεμλίνου. Ε, επιβάλαμε αυτές τις κυρώσεις ε, για το όσα έκανε η Ρωσία σε Ουκρανία και Κρυμνία πριν από πέντε χρόνια, αλλά σημάδια βελτίωσης δεν αναφέρονται. Αντιθέτως, είναι ακόμη περισσότερη η αυθαιρεσία στο εσωτερικό της Ρωσίας. Οπότε αυτός ο νόμος για τους ξένους πράκτορες μας δείχνει ότι υπάρχει γύρισμα στη χώρα και όχι πρόοδος όσον αφορά τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Με αυτό τον νόμο θίγονται όχι μόνο οι Ρώσοι. Αποτελεί αυτό ευθύ επίθεση κατά ημών των Ευρωπαίων αυτά που ενώνουν ξένους πράκτορες, αυτά που θεωρούν ε, βλαβερά, είμαστε εμείς πέραν των ακτιβιστών, έχουν στιγματιστεί και οι διπλωμάτες μας. Θα πρέπει να επιβάλλουμε και άλλες κυρώσεις πριν είναι αργά, να κάνουμε τη δουλειά μας ε, σε αυτούς που θέλουν να υπάρξει αυτός ο, αυτός ο νόμος Μαγνίτσκι. Αυτή είναι μια πολύ καλή εβδομάδα για την ελευθεροτυπία και την ελευθερία της έκφρασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη Δευτέρα στο Ευρωκοινοβούλιο λάβαμε την απόφαση να δημιουργήσουμε ένα βραβείο για τη βράβευση της ερευνητικής δημοσιογραφίας, καθώς και για τους καταγγέλλοντες και το σχετικό νόμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Τετάρτη τιμήσαμε την ελευθερία έκφρασης ενός Ουιγούρου. Αποδώσαμε απονείμαμε το βραβείο ε, το βραβείο Ζαχάροφ στον Ιλάν Τόχτη, ε, έναν από τους αντιφρονούντες ε, πανεπιστημιακό και διανοούμενο στην Κίνα. Όμως αυτό που συμβαίνει στην ε, Ρωσία είναι ανησυχητικό. Η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να διευρύνει το νόμο για τους ξένους πράκτορες και να καλύπτει αυτό και οι ιδιώτες, αυτό θα πλήξει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία στη χώρα. Θέλω να αναφέρω όλος ιδιαίτερος Το Radio Liberty, τη ραδιοφωνική υπηρεσία ειδήσεων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει δώσει πολλές ακριβείς και αντικειμενικές ειδήσει για τη Ρωσική Ομοσπονδία και τώρα αντιμετωπίζουν ε, πιέσεις. Ευχαριστούμε ο κύριος Μαριανή από την ε, ομάδα ID. Το ψήφισμα αυτό καταγγέλει ταυτόχρονα τη Ρωσία αλλά και τη ΣΥΠΑ. Να θυμίσω το 1938 ο νόμος Φάρα, ο οποίος σε πολλά σημεία θύμιζε αυτό που τώρα ψηφίζεται στη Ρωσία, καταδίκαζε τότε τους ξένου πράκτορες ε, στην Αμερική. Εδώ λοιπόν πρέπει να θυμηθούμε τις ε, εχθρότητε ε, που υπάρχουν στο παγκόσμιο προσκήνιο και καμιά φορά ξεπερνούν την κοινή λογική. Εδώ θα πρέπει να διατηρήσουμε τις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία αλλά χρειάζεται αυτό για τον νόμο των ξενοπρακτόρων, διότι αυτό βλάπτει και την ε, οικονομία μα. Ε, ε, όπου κάτι γίνεται, βλέπουμε από πίσω τον Πούτιν. Brexit, εκλογέ στη Γαλλία κτλ. Ε, εδώ λοιπόν θέλουμε αντίπεινα, θέλουμε να παγώσουμε τα ε, περιουσιακά των ολιγαρχών. Η Γαλλία προέβλεψε ένα νόμο το 1998 που δεν επιτρέπει σε ξένους να οργανώσουν και να συνασπιστούν στην επικράτεια της χώρας δικές τους, ε, δικούς τους οργανισμούς. Αυτό που πρέπει να κάνουμε με τη Ρωσία είναι να περάσουμε σε διάλογο και κάνουμε το αντίθετο, μπαίνουμε σε αδιέξοδο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κρασνοντεύσκε από τους Ιδρυτικούς και Μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πιο αυστηρή εκδοχή του νόμου για τους ξένους πράκτορες είναι ένα σύμπτωμα που δείχνει ότι η ρωσική κοινωνία θέλει να απομακρυνθεί από την πραγματική πληροφόρηση και τον έξω κόσμο. Είναι μια αντίδραση του καθεστώτος του Πούτιν απέναντι σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες όπου υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Nord Stream 2 ε, και ο σχετικός αγωγός και οι Ρώσοι αναγκάζονται να είναι ευχαριστημένοι με την ε, κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, ενώ θέλουν να διαμαρτυρηθούν για την οικονομία και τι συνθήκε διαβίωσή του. Υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα στη χώρα, κοινωνικά, οικονομικά και με και αυτά ε, ουσιαστικά καλύπτονται πίσω από μία ε, σωρία και εκφράσεων και παραμυθιών περί πολιορκούμενου ορχηρού. Πρέπει η Ρωσία να εκδημοκρατιστεί και θα πρέπει η Ρωσία ίδια να καθορίσει το, την πορεία της και να αποφασίσει ποια, ποιο δρόμο θέλει να πάρει. Ευχαριστούμε και τώρα ο κύριος Βίλουμσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ελευθερία της έκφρασης, το δικαίωμα του συνασπίζεστε, είναι ε, ακρογωνία η λύθη της Ευρωπαϊκής ε, Διακήρυξης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου έχει προσπογράψει και η Ρωσία. τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τα βασικότερα θεμελιώδη δικαιώματα, που εμεί θεωρούμε δεδομένα, να δέχονται πιέσεις. Τα πολιταρχικά καθεστώτα εργάζονται συστηματικά για να καταστρέψουν την κοινωνία των πολιτών. Το βλέπουμε εντός των δικών μας συνόρων, στην Ουγγαρία με τον Ορμπάν, στο Ισραήλ με τον Νετανιάχου ε, και βεβαίως και στη Ρωσία με τον Πούτιν. Ας είμαστε λοιπόν πολύ σαφείς σήμερα. Δεν δεχόμαστε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα να δέχονται επιθέσεις ή η κοινωνία των πολιτών να δέχεται πλήγματα. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε η ρωσική κυβέρνηση να μην εγγυάται ως οφείλει την ελευθερία του συνασπίζεστε, του οργανώνεστε και της έκφρασης. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ζαντατσόφσκι. Pokiaľ Európska únia chce existovať v takej podobe, ako existuje a chce sa hrať na sucu sveta... Ευχαριστώ, αλλά όπως βλέπουμε ως σήμερα η κατάσταση στη Ρωσία δεν αλλάζει. Εάν εμεί όμω θέλουμε να είμαστε και οι θεματοφύλακε των, αρχο... των ε, οικουμενικών αξιών παγκοσμίω, πρέπει να είμαστε και αντικειμενικοί. Εδώ δεν βασιζόμαστε σε πραγματικά γεγονότα και στοιχεία, ούτε είμαστε αντικειμενικοί στην κρίση μας. Η αντιπολίτευση στη Ρωσία δεν ξέρω εάν πραγματικά δέχεται τις πίεσεις που λέμε. Εγώ έχω κάνει τον κόπο να ασχοληθώ με όλου τους νόμους που έχω περάσει από, Ρωσική, από τη Ρωσική Βουλή από το 2012 μέχρι το 2015. Οι νόμοι αυτοί έχουν γίνει δεκτέ το 60% της ε, Ρωσικής Δούμας. Και οι, τα κόμματα τη αντιπολίτευση δεν καταψήφισαν του νόμου. Άρα είναι κάτι που δεν θέλει μόνο η κυβέρνηση τη Ρωσία, αλλά είναι απάντηση στα, αμερικανικέ κυρώσει. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και όχι να είμαστε ρωσόφοβοι. Ο κόσμο δεν μπορεί να γίνεται αντιληπτό μόνο μέσα από το δικό μα το βλέμμα. Ε, χρειαζόμαστε επίση ε, και συνεργάτε για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να χτίσουμε γέφυρε και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό πρέπει να κάνουμε και με τα άλλα κράτη. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ε, παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο αγόρευσης. Ο κύριος Λέγκα, επόμενος ομιλητής. Οι ε, χριστιανοδημοκράτες έχουν ως θεμέλιό τους την κοινωνία των πολιτών. Εγώ είμαι χριστιανοδημοκράτης και μια ισχυρή ε, ε κοινωνία ε, είναι αυτό που με ενδιαφέρει. Ο Πούτιν δεν ξέρει τι είναι η κοινωνία των πολιτών. Νομίζει ότι είναι απειλή ε, στο αυταρχικό του καθεστώς που διαρκεί και ε, έχει βάλει κάποια κουτάκια τα οποία κάθε φορά ε, χρησιμοποιεί και τσεκάρει. Εκφοβίζω τον τύπο τσεκ. Ε, και νόμος για τους ξένους πράκτορες τσεκ. Κερδίζω εκλογές τσεκ. Και πάλι προσπαθεί να αφημώσει την πολιτική αντιπολίτευση που κατά την άποψη του Πούτιν δεν θα πρέπει να υφίσταται. Αλλά υπάρχει και πρέπει να υπάρχει και όχι μόνο στη Ρωσία. Όσο και αν είναι πράκτορας, ε, πρώην πράκτορας της ΚΑΓΕΜΠΕ, ε, δεν υπάρχουν παντού ξένοι πράκτορες σε κάθε γωνία. Βλέπει μπροστά του παντού πράκτορες. Εγώ ε, είμαι στεναρός χριστιανοδημοκράτης και υποστηρίζω την κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστώ. Άρα κόβαρτς από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. πρέπει να πω ότι ε, και εγώ ε, έχω μιλήσει ε, για αυτό το θέμα και στο παρελθόν. Έχουμε εκφράσει ε, την αλληλεγγύη μας προς τον ηγέτη των Ουιγούρων αυτή την εβδομάδα, τον Ιλάμ Τότι, που αγωνίζεται κατά της, της κυβέρνησης της Κίνας. Και τώρα ασχολούμαστε με τη Ρωσία και τον περίφημο νόμο ε, ο οποίος θέλει να χαρακτηρίσει ε, ξένους πράκτορους ο οποίος ε, διαφωνεί με την κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν αντιφρονούντες, όλοι είναι ξένοι πράκτορες. Δεν θα μπω σε υπερβολικές αναλύσεις. Ξέρουμε τι καθεστώς είναι αυτό το Πούτιν. Δεν θέλει απλώς να περιορίζει και να φημώνει τον κόσμο στη χώρα του, αλλά εξάγει και το προϊόν αυτό. αυτή την καταστολή και πραγματικά λυπάμαι για την εξαγωγή ε, της καταστολής και στην ίδια μου τη χώρα που έπεσε το πρώτο θύμα σε αυτό το βωμό. Είναι πολύ μεγάλο κρίμα. Σήμερα στην Ουγγαρία η κοινωνία των πολιτών ε, είναι ε, πάρα πολύ τραυματισμένη, χωλαίνει κυριολεκτικά ε, προσπαθούν να καταργήσουν όλες αυτές τις δομές. Είδατε τι έγινε με το Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Ευρώπης. Δεν ξέρω εάν γνωρίζετε ε, από ποια κονδύλια προέρχονται ε, αυτές οι χρηματοδοτήσεις. Είναι από τους δικούς σας φορολογουμένους. Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Ντονάτα από το Ευχαριστώ. Πρέπει να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Όχι μόνο γιατί υπάρχει καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί, αλλά και γιατί η ρωσική μαφία δεν σταματά στα ρωσικά σύνορα. Το έχω ήδη επισημάνει ότι η παραπληροφόρηση που πηγάζει από τη Ρωσία απειλεί εκ των έσω την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα ε, και στη Ρωσία και στην Ουγγαρία η, αντιφο, η αντιπολίτευση, οι πολιτικοί αντίπαλοι, οι δημοσιογράφοι είναι στο στόχαστρο και μάλιστα και στην Ουγγαρία δοκιμάζονται ρωσικές μέθοδοι. Και μάλιστα έχουμε μία ολόκληρη ρωσική ομάδα κατασκόπων που έχουν εγκατασταθεί στην Ουγγαρία και προσπαθούν να επηρεάσουν τα ουγγρικά μέσα μεζική ενημέρωση, φιλτράροντα ανακριβεί ε, και φαλκιδευμένε ειδήσει. Θα πρέπει να προστατεύσουμε το ελεύθερο πνεύμα των ΜΚΟ και να μην επιτρέψουμε την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του στη Ρωσία. Κύριε Ρόμπετ, χθε απονείμαμε το βραβείο Ζαχάροφ ε, στον Ήλαμ Τότι και ε, είχαμε και δύο πολύ σημαντικούς φιναλίστες υποψηφίους για το βραβείο αυτό. Και τώρα συζητούμε το ρωσικό νόμο για τους ξένους πράκτορες που απειλεί τις ΜΚΟ και τους δημοσιογράφους. Αυτό δείχνει δύο όψεις ε, αυτού του νομίσματος ε, της προσπάθειας υπόσκαψης των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των χωρών που δεν έχουν την τύχη να ανήκουν σε αυτή τη Συμμαχία Ελεύθερων Εθνών. Ε, εγώ παρακολούθησα αυτό το θέμα, μια εποχή μάλιστα που η ελευθερία έκφρασης και λόγου ε, απειλείται όλο και περισσότερο αυτό το πιο πολύτιμο αγαθό που έχουμε. Μάλιστα χθες ε, είδα ότι απουσίασαν ε, από την τελετή απονομής του βραβείου Ζαχάροφ τα μέλη του κόμματος Brexit. Και πάλι ο Μπόρις Τζόνσον βρήκε νέους τρόπους για να καθυστερήσει τη δημοσίευση της έκθεσης για την ρωσική παρέμβαση στις βρετανικές εκλογές. Αυτά και δεν θα ήθελα να πω τίποτα άλλο. Ο κύριος Στέρτς τώρα έχει το λόγο από το ECR. Καλημέρα σας. Ε, καλημέρα, Πρόεδρε. Τα νέα μέτρα του Κρεμλίνου περιορίζουν ακόμα περισσότερο τις ελευθερίες των Ρώσων πολιτών και όλων των ανεξαρτήτων οργανώσεων. Ε, οι νόμοι του 12 και του 15 για τους ξένους πράκτορες πέτρεψαν να διωχθεί οποιαδήποτε οργάνωση που έχει σχέση με το εξωτερικό και τις οποίες οι δραστηριότητες δεν άρεσαν στην εξουσία. Με τους νέους κανόνες κανένας δεν μπορεί να έχει στη Ρωσία επαφές με το εξωτερικό που να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν διοικητικά ή ποινικά εναντίον του. Πολύ μοιάζουν όλα αυτά με την, με την Σοβιετική Ένωση και την κομμουνιστική δικτατορία πριν από το 1985 όταν έφτασε η Περιστρόικα και ο Γκρομπατσόφ. Είναι τραγική αυτή η αντιδημοκρατική εξέλιξη που μάλιστα παραβιάζει όλες τις δεσμεύσεις της Ρωσίας στο διεθνές επίπεδο ε, και στις συνθήκες. Γι' αυτό ζητάμε από τον πρόεδρο Πούτιν να μην καταδικάσει τη Ρωσία ακόμη περισσότερο σε αυτή την ε, οπισθοδρόμηση που της επιβάλλει η απομόνωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Fox τώρα είναι πολύ επικίνδυνη ε, απειλή στην ελευθεροτυπία και δείχνει την ξενοφοβία στη Ρωσία. Όμως έχω ακούσει τόσο πολλές συζητήσει σε αυτή την αίθουσα που πολύ εύκολα κατα... Ε, κατηγορούν τις ξένες παρεμβάσεις για όλα. Ε, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έχει το ηθικό κύρος για να επικρίνει τη Ρωσία, καλύτερα είναι να καθαρίσει τα του οίκου της πρώτα. Πόσες φορές εδώ έχουμε ακούσει ευρωβουλευτές, επιτρόπους και εργατικούς που δεν συμμορφώνονται προς την Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκή ατζέντα ότι είναι ξένοι πράκτορες του Πούτιν, οι Ρώσοι, ε, ε, ρωσικοί δάκτυλοι που ελέγχουν ε, τα πράγματα ή που παρεμβαίνουν, ας πούμε, όπως το ε, δημοψήφισμα για το Brexit. Οι καταδίκες και οι κατηγορίες για εξωτερική συνεργασία δείχνουν ξενοφοβία στις ίδιες μας τις χώρες. Επίσης, θεωρούν πως οι ψηφοφόροι μας είναι, δεν έχουν την ικανότητα να κρίνουν μόνοι τους εφόσον διαρκώς κατηγορούμε τους ξένους ότι επηρεάζουν. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε διαρκώς τους άλλους. Θα πρέπει να είμαστε ακατάβλητοι στο να επικρίνουμε την ε, ε, τον τρόπο του Πούτιν να περιορίζει τον ίδιο του το λαό. Αλλά το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και εδώ. Δεν πρέπει να ε, διαρκώς να κατηγορούμε τους ξένους για τις δικές μας αποτυχίες. Προσοχή να προσέχουμε τα του οίκου μας. Ευχαριστώ πολύ κύριο Σέλ για το... ο κύριος Κέλ για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ ο Ρωσικό νόμο για του ξένου πράκτορες είναι πολύ ανησυχητική εξέλιξη για την ελευθερία της ρωσική κοινωνία και τη ελευθεροτυπίας στη Ρωσία. Δημιουργείται ένα εχθρικό περιβάλλον, όλο και πιο εχθρικό για του δημοσιογράφου, Επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα στι ΜΚΟ, στου δημοσιογράφου που αντιμετωπίζουν προβλήματα μεγαλύτερη καταστολή ενώ προσπαθούν ουσιαστικά ε, να προωθήσουν ε, την ε, πληροφόρηση. Στιγματίζονται οι δημοσιογράφοι Γράφει ως ε, ξένοι πράκτορες. Ε, είναι κακό για τη δημοκρατία και πρέπει να το καταδικάσουμε ε, σε ένα περιβάλλον που οι ελευθερίες συρρυκνούνται. Και πραγματικά ουσιαστικά είναι ένα μέσο εκφοβισμού αυτό ο νόμο για να φημώσει του δημοσιογράφου και τη ΜΚΟ. Πρέπει να καλέσουμε τι ρωσικέ αρχέ να ευθυγραμμίσουν την νομοθεσία του με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα παγκόσμια πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο από την ομάδα των σοσιαλιστών από τη Σοσιαλική Μαγιορίνου. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ελευθεροτυπία και η ελεύθερη ενημέρωση είναι ουσιαστικά στοιχεία για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Όμως ο Βλαδιμίρ Πούτιν παριστάνει πως δεν το γνωρίζει και προσπαθεί μέσω νέων νόμων να μπορεί να πάρει χρηματοδοτήσει για οργανώσεις που δεν είναι ευπρόσδεκτε γιατί θεωρούν, θεωρούνται ε, ε, ξένοι πράκτορε Και έτσι φτιάχνει ένα κατάλογο που προελιότερα αφορούσε του ΜΚΟ και διάφορες ξένες οργανώσεις και τώρα και τα blog. Είναι προφανές ότι, είναι, ε, ότι βλέπουμε μία μανιακή κατάσταση, μία έμονη ιδέα να ελέγξει την πληροφόρηση και να περιορίσει οποιαδήποτε απόκληση. Και σωστό είναι να το καταδικάσουμε εδώ όπως το κάνουμε, αλλά θα πρέπει να το σκεφτούμε και να σκεφτούμε τους φίλους του Πούτιν, οι οποίοι είναι μεταξύ μας και να σκεφτούμε αυτό το ε, ε, σχέδιο σχέδιο που είναι ένα κοινωνικό σχέδιο διότι ε, δεν μπορούμε να το δεχτούμε διότι είναι αντίθετο με τις αξίες μας και τη δημοκρατία μας. Ο κύριος Μπένιον από το Ρινιού είναι ο επόμενος ομιλητής. Thank you, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, η αναθεώρηση τη ομοθεσία θα επιτρέψει στη ρωσική κυβέρνηση ανεξάρτητου δημοσιογράφου και συντάκτε στο λονιό που παίρνουν χρηματοδότηση από οποιαδήποτε ξένη πηγή να του θεωρεί ή να του ονομάζει ξένου πράκτορε, που ουσιαστικά σημαίνει πολιτικό αντιφρονών. Και θα πρέπει τελικά να βάζουν ετικέτε στο έργο του, ε, να αντιμετωπίζουν αλλιώ πρόστιμα ή και φυλακή μέχρι δύο έτη. Ο νόμο αυτό ουσιαστικά θα φημώσει την κριτική κατά τη κυβέρνηση, προστατεύοντα περισσότερο την ελευθεροτυπία, την ανεξαρτησία των μέσων, ε, την ελευθερία τη έκφραση. Καλό τη ρωσική κυβέρνηση να, να κρούσει πρίμναν ε, και να ευθυγραμμίσει την νομοθεσία τη με τι υποχρεώσει ε, που έχει δυνάμει του διεθνού δικαίου και να πάψει να προσπαθεί να καταστέλει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία και την κοινωνία των πολιτών. Είναι λυπηρό να ακολουθεί η Ρωσία αυτή την προσέγγιση όσο μάλιστα βλέπουμε ότι μπαίνει ξανά στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ροπέ, εκ μέρους των Πρασίνων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η μεγαλύτερη απειλή για το κρεβλίνο είναι η δημοκρατία. Γι' αυτό και η Ρασία αναλαμβάνει δράση κατά των μη κυβερνητικών οργανώσεων και κατά του ελεύθερου τύπου και των πολυφωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που είναι οι μόνες πηγές αξιόπιστων και έγκυρων πληροφοριών. Και πραγματικά ακόμη και αυτούς που δίνουν μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την περιβαλλοντική προστασία που προσπαθούν να προσπίσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες βρίσκονται στο στόχαστρο του Κρεμλίνου προπαγανδιστική μηχανή του Πούτι βέβαια δεν έχει αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα για αυτόν και το καθεστώς αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή κρίση με δύο απειλές, μια εσωτερική και μια εξωτερική. Προσπαθεί να επέβει σε εκλογικές διαδικασίες και δημοψηφίσματα σε άλλες χώρες, αλλά γίνεται αυτό όλο και πιο δύσκολο για τη Ρωσία. Και βοηθώντας το ρωσικό λαό, νομίζω ότι δίνουμε μία διέξοδο στη λαχτάρα του για δημοκρατία και επιβίωση. κυρία Σόιντροβα, σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θυμάμαι ακόμη πολύ καλά τι σήμαινε όρος «ξένος πράκτορας» στην πρώην ε, Σοβιετική Τσεχοσλοβακία και το Ανατολικό Μπλοκ που βρίσκονταν υπό το ζυγό της Σοβιετικής δικτατορίας οι ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ζεχοσλοβακία τότε είχαν ε, υποστεί καταπίεση. Και τώρα έχουμε το Ρωσικό Υπουργείο Δικαιοσύνης που χρησιμοποιεί τον όρο «ξένος πράκτορας» για να καταδιώξει ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ακόμη και ιδιώτες. Μάλιστα, μέσα στις οργανώσεις που βρίσκονται στο στόχαστρο βρίσκεται και μια τσεχική οργάνωση. Οι άνθρωποι ε, που έχουν ανάγκη. People in need. Επίσης, ανθρωπιστικές οργανώσεις ε, που ασχολούνται με αναπτυξιακή βοήθεια στον τρίτο κόσμο βρίσκονται και αυτές στο κατάλογο. Άνθρωποι και οργανώσεις που προστατεύουν ε, τα δικαιώματα της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία, αντιφρονούντες, πολιτικοί αντίπαλοι, είναι όλοι θύματα καταδίωξης. Ακόμη και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που δεν λαμβάνουν δηλαδή καμία εξωτερική χρηματοδότηση, αντιμετωπίζονται ως ανεπιθύμητοι ξένοι πράκτορες. Νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε κατάργηση αυτού του νόμου. Στρουγκάριου από την ομάδα Ρινιού. Ευχαριστώ. Το ε, ραδιόφωνο Ελεύθερη Ευρώπη ε, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη επί Σοβιετικής Ένωσης και είχε μπει στο, στη μαύρη λίστα μαζί με, άλλες, ε, ε, με άλλους ελεύθερους ε, σταθμούς. Μάλιστα ο νέος νόμος, ο συγκεκριμένος νόμος για τους ξένους πράκτορες είχε πρωτοεγκριθεί το 2012 υποχρεώνοντας εγγραφή στο Μητρό ΜΚΟ και σταθμό που λάμβαναν ε, εξωτερική χρηματοδότηση. Τώρα επεκτάθηκε αυτό ο νόμο, ε, διευρύθηκε το πεδίο του και περιλαμβάνει ακόμη και ιδιώτε, δημοσιογράφου ή πολιτικού αντιπάλου, χαρακτηρίζοντά του ξένου ε, πράκτοτε. Είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα η πολιτικου αντιπαλου χαρακτηριζοντα του ξενου πρακτορες πολυφωνία των ΜΜΕ και καταπιέζεται βάναυσα από την ρωσική κυβέρνηση. Θα πρέπει να ζητήσουμε κατάργηση αυτού του νόμου που παραβιάζει την ελευθερία έκφραση και λόγου και τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφέ. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, μία εξομάλυση στο σχέσιο με τη Ρωσία εφόσον καταπατά περίτρανα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Πούτιν δεν σέβεται τίποτα. Θα πρέπει να υιοθετήσουμε ένα αντίστοιχο νόμο με αυτό του Μαγνίτσκι. Ευχαριστώ πολύ. Έχω εννέα αιτήσει ε, για τη διαδικασία προσέλκυση της προσοχής του Πρόεδρου. Σε έξι μόνο μπορώ να δώσω το λόγο. διονόμαδα ομάδα. από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, για οποιονδήποτε μπορεί να έχει κάποιε αμφιβολίες για το κατά πόσο ο Πούτιν είναι δικτάτορας ή όχι. Έχετε πλέον ε, την απάντηση, έτσι δεν είναι με αυτό το νόμο. Τόματς, ε, είναι Εύκολα μπορεί κανείς να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται ουσιαστικά για τη δίωξη ε, ανθρώπων που προσπαθούν να προωθήσουν τη δημοκρατία, την ελευθεροτυπία, την ελευθερία έκφραση, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, πραγματικά αυτό που συμβαίνει ε, πρέπει να μας ανησυχήσει. Είναι ένα σκόδανα συναγερμού για τους ηγέτες της κοινή γνώμης, η ρωσική αντιπολίτευση, οι δημοσιογράφοι, όλοι αντιφρονούντες διώκονται από τον Πούτιν. Παρακαλώ λοιπόν τον το εκπρόσωπο κάτι να κάνει ε, για να υπερασπιστούμε τα εκατομμύρια Ρώσ πολίτες ε, που ε, θέλουν να στραφούν στην Ένωση με ελπίδα. Πρόεδρος. Λόπεθ Αγγιλάρου, επόμενο Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, κύριε Πατεκπρόσωπο Μπορέλ, το ψήφισμα που θα ψηφίσουμε για τον ρωσικό νόμο περί ξένων πρακτόρων στο Κοινοβούλιο περιλαμβάνει δύο προτεραιότητε. Πρώτον, πρόσβαση στην ελεύθερη πληροφόρηση και την ελευθερωτική ε, Δάφνη Καρουάνα και ε, βραβείο Ζαχαφ. Δεύτερον, όμω, παρέμβαση τη Ρωσία και στα, στα σύνορα αλλά και εκτό στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι ένας χώρος ειρήνης, ε, γι' αυτό υπερηφανεύεται. Υπήρξαν όμως ε, κάποιες ε, πραγματικά εχθρικές πράξεις κατά της Γεωργίας, της Ουκρανίας, της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν από τη Ρωσία. Μιλάμε για τα σύνορα της πρώην Σοβιτικής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν η παρέμβαση της Ρωσίας να μας ανησυχεί. Μιλάω για παρέμβαση στον κυβερνοχώρο. Πρέπει απερίφραστα να καταδικάσουμε όλες αυτές τις ενέργειες, τις επιθέσεις κατά δημοσιογράφων, συντακτών ιστολογίων και άλλων, κατά ενός καθεστώτος που τα ελέγχει όλα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Γκουε τώρα, η κυρία Αντάλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το 2017, όταν ε, ήταν στο αποκορύφωμά της ε, η ρωσική παρέμβαση, ζητήσαμε να καταγραφούν οι ξένοι πράκτορες υπό το νομοσχέδιο καταγραφής των ξένων πρακτόρων. Ήταν προφανές ότι η Ρωσία θα έκανε και τα αντίστοιχα. Είναι βασική αρχή των διεθνών σχέσεων. Κάθε ενέργεια έχει και το αντίθετό της και η Ρωσία ακριβώ αυτό κάνει. Δυστυχώς μάλλον θα επιβληθεί αυθαίρετα, θα είναι εις βάρος των ανεξαρτήτων δημοσιογράφων και των οργανώσεων των πολιτών στη Ρωσία. Αρκεί θα δούμε τι, έχει κάνει, τι έχουν κάνει οι Ηνωμένε Πολιτείε με το δικό τους νόμο περί, εξων, ε, περί ξένων πρακτόρων. Η, Μαρία που Πουτίνα βρίσκεται σε, κατηγορείται μάλλον πράκτος απλά και μόνο επειδή είναι Ρωσίδα. Οι Ρώσοι στην ουσία αντιγράφουν αυτά που κάνουν άλλοι στην Δύση. Μόλις το σταματήσουμε αυτό και πάψουμε να, να χρησιμοποιούμε τους Ρώσους ως σκιάχτρο θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Ο κύριος Ποσπίσιλ του ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ. Αυτή η νομοθεσία αποδεικνύει ότι το ρωσικό καθεστώς ε, καθίσταται διαρκώς πιο ε, αυταρχικό. Εμεί στην Τσεχία γνωρίζουμε περί τίνο πρόκειται. Έχουμε έναν πρόεδρο, τον κύριο Ζέμαν, που μάλιστα υποστηρίζει το καθεστώ του Πούτιν. Εμεί όμω οφείλουμε να διαμαρτυρηθούμε και χαίρομαι για το γεγονό ότι με αυτό το ψήφισμα, το οποίο υποστηρίχθηκε και από το πνεύμα της προηγούμενης νομοθεσίας, σχετικής νομοθεσίας καταδικάζει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ρωσική Ομοσπονδία. Καταδικάζουμε επίσης κάθε παρέμβαση των ρωσικών αρχών στις δικές μας χώρες και την παρέμβασή τους στις προεκλογικές εκστρατείες. Η Ρωσία θα πρέπει να είναι εταίρος μας, ναι, αλλά όχι η Ρωσία του Πούτιν. Και αυτό πρέπει να το πούμε ε, καθαρά και εξάστερα από πλευρά της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να επιτρέπει τέτοιο ε, προπαγάνδα από πλευρά του ρωσικού καθεστώτος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γραπίνη, έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Η πρώην Σοβιτική Ένωση ήταν, ε, είναι καταπιεστική, ε, άτεκτη, αμήλικτη. Ε, και εμείς από το πρώην Ανατολικό Μπλοκ ε, έχουμε βιώσει το πετσί μας τέτοιου είδους παραβιάσεις. Καταδικάζουμε το νόμο που πρόσφατα έχει αναθεωρηθεί με διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή τους. Ποτέ δεν θα μάθουμε την αλήθεια αν καταπιέζονται συστηματικά οι μόνες έγκυρες και αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης. Η κοινωνία της Ρωσίας θέλει ελευθερία έκφρασης και λόγου, θέλει δημοκρατία. Φυσικά και θα υπερψηφίσουμε το ψήφισμα. Είμαστε γείτονε τη Ρωσία, αλλά θα πρέπει να ενισχύσουμε το σεβασμό των δημοκρατικών κανόνων. Μόνο έτσι θα γίνουμε καλή εταίροι. Και τελευταίος ομιλητή στη διαδικασία Κατσδιά, κυρία Μόλτι. Σας ευχαριστώ. Ως Είχαμε την ε, Ρωσία γείτονα και τα έχω ζήσει τα πράγματα και πρέπει να σας πω ότι πάντοτε υπήρχαν φιλικές σχέσεις, ε, υπήρχαν ε, ανταλλαγές με αυτή τη χώρα. Τώρα όμως οι διάφορες οργανώσεις δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Η κοινωνία των πολιτών έχει φημωθεί και καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται για μια σημαντική απειλή. Ο νόμος το μόνο που κάνει είναι να επιδεινώνει την κατάσταση γιατί οι ελευθερίες συρρυκνούνται όλο και περισσότερο. Δεν μπορούμε λοιπόν να ανεχθούμε τη θυμόση και τις αντιπολίτευσης, γιατί εδώ μιλάμε πλέον για δικτατορία. Ήδη ο επικριτικός τύπος φημώθηκε, οι δημοσιογράφοι ε, όπως η Άννα για ε, διώκονται και έχουν χάσει μάλιστα και τη ζωή τους όπως η Πολιτόσκαγια και άλλοι δημοσιογράφοι ε, και θα πρέπει με την ε, αντιπολίτευση και την κοινωνία των να αγωνιστούμε. Σε... Ωραία, ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο. Το λόγο έχει ο ύπατος εκπρόσωπος, ε, ο κύριος Μπορέλ, για να ολοκληρώσουμε και τη συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σαφέστατη και μακροχρόνια στάση για το νόμο της Ρωσίας και τους ξένους πράκτορες. Και η τελευταία αναθεώρηση αυτού του νόμου που υπεγράφει από τον πρόεδρο Πούτιν στις 2 Δεκεμβρίου επεκτείνει το σημείο, το πεδίο εφαρμογή του νόμου για τους ξένους πράκτορες προκειμένου να περιλαμβάνει και ιδιώτες. Και πολλοί από εσά ε, εκφράσετε τις έντονες ανησυχίες σας για αυτή την επέκταση του πεδίου εφαρμογή και δικαίως εύλογα γιατί ε, έτσι μπορεί να επηρεαστούν δυνητικά ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, συντάκτες ιστολογίων, bloggers και είναι ένα επιπλέον βήμα για τον περιορισμό της ε, πολυφωνίας του ΜΜΕ, της ελευθερίας έκφρασης και του λόγου στην Ρωσία. Από το 2012, όταν πρωτοεγκρίθηκε ο νόμος για τους ξένους πράκτορες στη Ρωσία, έδινε τη δυνατότητα σε ΜΚΟ να χαρακτηρίζονται ξένοι πράκτορες. Πάνω από 150 ΜΚΟ έφεραν αυτό το στίγμα, αυτή την ταμπέλα στον στον τίτλο τους. Οπότε ε, πρέπει να υποστούν αυτό το στιγματισμό και να ε, υποβληθούν σε ελέγχους και επιθεωρήσεις και αυτός ο περιορισμός των θεμελιωδών ε, ε, ελευθεριών περιόριζε τους ήδη πενιχρούς πόρους χρηματοδότησης του ΜΚΟ και αποδυνάμωνε την κοινωνία των πολιτών στη Ρωσία. Μάλιστα το 2017 ο σχετικός νόμος για τους ξένους πράκτορες επεκτάθηκε ακόμη περισσότερο σε οποιαδήποτε ΜΜΕ που ελάμβανε ξένη χρηματοδότηση άμεσα ή έμεσα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ξένος πράκτορας. Οπότε συρρυκνώθηκε ακόμη περισσότερο ο χώρος για τα ελεύθερα και ανεξάρτητα ΜΜΕ και για τις ανεξάρτητες φωνές στη Ρωσία. Ο νόμος για τους ξένους πράκτορες αντιβαίνει στις υποχρεώσεις της Ρωσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επανειλημμένως έχει καταδικάσει αυτή την νομοθεσία και μάλιστα πολύ πρόσφατα σε μία δήλωση Τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τον εκπρόσωπο της ΕΙΕΔ στις, 30, 23 ε, Νοεμβρίου. Καταδικάσαμε ε, αυτό το νόμο και μάλιστα η επέκταση του πεδίου εφαρμογή περαιτέρω διεύρυνση είναι ακόμη μια χειρονομία και κίνηση περαιτέρω συρρήκνωση και περιορισμού τη ελευθερία έκφραση. Ζητούμε από τι ρωσικέ αρχέ να σεβαστούν τι διεθνεί του υποχρεώσει για την ελευθερία του συνέρχεστε, του συνεταιρίζεστε και την ελευθερία λόγου και έκφραση. Ε, είναι ζωτική σημασία να δίνονται οι Ευρωπαίοι πολίτε να ασκήσουν αυτά τα δικαιώματα του συνέρχεστε, του, συνεταιρίζεστε ή τη συμμετοχή σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις που προωθούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και την κοινωνία των πολιτών στη Ρωσία. Είναι κάτι που κάνουμε άλλωστε παντού, γιατί αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η δική υποστήριξη είναι σημαντική και καλό είναι να κάνουμε δημόσιες δηλώσεις, να συμμετέχουμε για να παρακολουθούμε δίκες ε, και να έχουμε συνεχείς επαφές με την κοινωνία των πολιτών. Παρακολουθούμε εκ του σύνεγγε της εξέλιξη στη Ρωσία και ζητούμε από τις αρμόδιες αρχές να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους και τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο ίδιο το Ρωσικό Σύνταγμα. Επίση, επιμένουμε στην ανάγκη να γίνουν σεβαστέ οι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και γενικώ ε, οι συμβάσει του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως κατοχυρώνονται σε αυτές τις συμβάσεις ε, ε, θα πρέπει να τηρηθούν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους Ευρωβουλευτές. Nagyon szépen köszönöm ezzel a vitát, lezárom. A vita lezárásához hat állásfoglalási indítványt kaptam. Σας ευχαριστώ. Έχω λάβει ψηφί... Ε, ε, ε, ψηφίσματα. Μετά από λίγα λεπτά στις 12 ακριβώς θα ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες. Yeah.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε μια απόφαση ε, στην υπόθεση σε 502-2019 Γιουνκέρας και Βίας. Είναι μια απόφαση εξαιρετικά σημαντική που αφορά ακριβώς την σύσταση του σώματος. Δεν χαζολογούσαμε και να σας κάνουμε να περιμένετε έτσι χωρίς λόγο. Το δικαστήριο λοιπόν αποφάσισε ότι η ανάληψη της κοινοβουλευτική εντολής προκύπτει από την ψήφο των ψηφοφόρων. Το δικαστήριο λοιπόν δήλωσε ότι ένας άνθρωπος το οποίο η εκλογή στο Ευρωκοινοβούλιο επισήμως ε, έχει αναγνωριστεί από την αρμόδια αρχή του οικίου κράτους μέλους όπου έγιναν οι εκλογές από εκείνη τη στιγμή αποκτά την ιδιότητα του βουλευτή και χέρι της ε, κοινοβουλευτικής ασυλίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού που αφορά τα προνόμια και την ασυλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. του κανονισμού λοιπόν που αφορά τα προνόμια και την ασυλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη στιγμή της ανακοίνωσης των επισήμων αποτελεσμάτων. Κατά συνέπεια, μέλος του Ευρωκοινοβουλίου θα πρέπει να ε, θεωρείται κανείς από τη στιγμή που έχουν ανακοινωθεί τα εν λόγω αποτελέσματα. Μάλιστα το δικαστήριο δηλώνει ότι η ασυλία σημαίνει ότι τα μέτρα της ε, ε, προληπτικής ε, ε, προστασίας θα πρέπει να ε, ισχύει μέχρι ότου το εν λόγω μέλος έρθει στο Κοινοβούλιο και να λάβει καθήκοντα. Δηλαδή, σε περίπτωση που οι αρμόδιες εθνικές αρχές θεωρούν πως μια τέτοια, ένα τέτοιο μέτρο θα πρέπει να διατηρηθεί αφού το εν λόγω άτομο έχει αναλάβει καθήκοντα ως ε, Ευρωβουλευτής, οφείλει να ζητήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα από το Ευρωκοινοβούλιο την αναστολή της ασυλίας, την άρση της ασυλίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ε, κανονισμού. Κάνω έκκληση λοιπόν στις αρμόδιες ισπανικές αρχές για να τις καλέσω να ε, συμμορφωθούν προς την απόφαση αυτή και έδωσα εντολή στις υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου να ε, εξετάσουν όσο γίνεται πιο σύντομα την εφαρμογή των επιπτώσεων αυτής της απόφασης για την σύσταση του Κοινοβουλίου μας. Σας ενημερώνω ότι δεν θα δεχτώ ε, επικλήσεις στον κανονισμό για αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Um, Συνάδελφοι, μετά από αυτή τη σαφέστατη δήλωση του Προέδρου, δεν ε, χρειάζεται να ε, αρχίσουμε με διαδικαστικά για αυτό το θέμα. Θα ήθελα να καλωσορίσω την αντιπροσωπεία του Ουκρανικού Κοινοβουλίου που συμμετείχε στην ε, δέκατη Σύνοδο της Επιτροπής Σύνδεσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ουκρανία εχθές. Ε, Πρόκειται για μια σημαντική συνεδρίαση που ήταν η πρώτη που έγινε από την έναρξη της νέας νομοθετικής περίοδου τόσο για το Ευρωκοινοβούλιο όσο και για την Φερχόφνα Ράντα, το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας. Και γι' αυτό ήταν μια πολύ καλή στιγμή για να εξετάσουμε με φιλοδοξία και όραμα τα όσα προσπαθούμε να επιτύχουμε από κοινού. Αγαπητοί Ουκρανοί φίλοι, η πολύπλευρη και εντατική συνεργασία μεταξύ των κοινοβουλίων μας είναι το σύμβολο των κοινών μας δεσμεύσεων προς το ευρωπαϊκό μονοπάτι που ακολουθεί θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε αυτή την εβδομάδα στο Κοινοβούλιο και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην εργασία σας ως ε, βουλευτών στο μέτωπο της ενίσχυσης και της εμβάθυνσης της δημοκρατίας σας. Περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Να περάσουμε λοιπόν στι προτάσει σε ψηφίσματο ε, επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρώτον, Μπουρκίνα Φάσο, τροπολογία 2, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε στο ψήσμα για το Αφγανιστάν και συγκεκριμένα τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση αγοριών στην επαρχία Λόγκαρ. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 1, ονομαστικά, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται με πολύ μικρή διαφορά ψήφων. Λίγο γρήγορα έκρινα τα πράγματα. Προχωρούμε στην τροπολογία 1, ψήφι Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2, ψήφι Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 3, ψήφι κατά αποχές απορρίπτεται και το σύνολο του ψηφίσματος ψήφι υπέρ κατά αποχές το ψήφισμα για το Αφγανιστάν εγκρίνεται. Προχωρούμε στο επόμενο ψήφισμα για το ρωσικό νόμο περί ξένων πρακτόρων. Έχουμε μια ονομαστική ψηφοφορία της παραγράφου 13 του αρχικού κειμένου. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε του συνόλου του ψηφίσματος ψήφι περ, κατά, αποχές. Το ψήφισμα εγκρίνεται. Και τώρα ερχόμαστε στο ψήφισμα για τον εορτασμό της 30ης απαιτίου της Ρωμανικής Επανάστασης του Δεκεμβρίου 1989 ονομαστικά, με ονομαστική κλίση θα ψηφίσουμε το σύνολο του ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και προχωρούμε στο επόμενο ψήφισμα. We will now vote κατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα. Ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο παραγράφου 1 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και το τρίτο τμήμα με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 1, ψήφι κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, το ψήφισμα για την κατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα εγκρίνεται. Uh, Ωραία, οπότε περνάμε στο ψήφισμα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της Δημοκρατίας στην Ικαράγουα και ψηφίζουμε την παράγραφο 7 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ολόκληρο το ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και το τελευταίο μας ψήφισμα για τη βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν. Μετά την παραγραφό 1, τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την παράγραφο 7 του αρχικού κειμένου με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Μετά την παράγραφο 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική σκέψη G, τροπολογία 1, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε ολόκληρο το ψήφισμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτό και σας εύχομαι ειρηνικά Χριστούγεννα και ραντεβού με το νέο έτος. Περνάμε τώρα στις αιτιολογήσεις ψήφου. Σας δίνω μισό λεπτό για να εγκαταλείψετε αθόρυβα και ειρηνικά την αίθουσα για να μπορέσουν οι συνάδελφοι να μιλήσουν και να ακουστούν. so i'd now like to open the floor for uh, explanations of votes on. Περνάμε τώρα στις αιτιολογήσεις ψήφου. Πρώτα το ψήφισμα για τον εορτασμό της 30ης επαιτίου της ε, Ρουμανικής Επανάστασης του Δεκεμβρίου του 1989. Ο Ντάνιελ Χάναν έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είχα το προνόμιο ε, να βρεθώ στο Βουκουρέστι. ήμουν 18 χρονών και παρακολούθησα από πρώτο χέρι την Επανάσταση. Και μάλιστα ε, ήμουν σε ένα μπαρ που ήταν το μόνο μέρος που μπορούσε κανείς να παραγγείλει μπύρα. Γιατί μόνο ιταλικό βερμούθ και ένα άλλο λικέρ μπορούσε να τον αγοράσει κανείς στη Ρουμανία. Και ήταν πραγματικά ε, τρομερές εθισίες που γίνονταν από τη Ρουμανία τότε. Και θα πρέπει να θυμηθούμε ότι η Επανάσταση όχι μόνο στη Ρουμανία και σε άλλους σοβιετικούς δορυφόρους σήμαιναν το τέλος της ε, κατοχής και την αποκατάσταση της ε, κυριαρχίας. Εντάξει, δημοκρατία, φυσικά και ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά είχαν αντιληφθεί οι λαοί στις χώρες αυτές ότι δεν είχαν νόημα όλα αυτά αν δεν υπήρχε λογοδοσία από τους κυβερνώντες. Γι' αυτό και ο Σάλ είχε πει νωρίτερα ότι η εθνική κυριαρχία και η δημοκρατία ουσιαστικά είναι έννοιες που ταυτίζονται. Ευχαριστώ κύριε Χάναν. Ο κύριος ε, Άγγελ Τζαμπάτσκι έχει το λόγο. Ένα λεπτό μην ξεχνάτε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, όπως και ο κύριος Χάναν, παρακολούθησα και εγώ τα γεγονότα στην ε, Ρουμανία από την τηλεόραση και μάλιστα ε, εγώ ήμουν στη Σόφια πολύ κοντά δηλαδή στη Ρουμανία και βλέπαμε τι γινόταν στους δρόμους της Μισοάρα και σε άλλες ρουμανικές πόλεις. Τότε ε, η Ρουμανία βρισκόταν στο έλεος μιας κομμουνιστικής δικτατορίας που προσπάθησε να καταστρέψει τη μνήμη των λαών μας και την αυτοδιάθεσή μας. Μια δικτατορία που προσπάθησε να δημιουργήσει ένα νέο είδος πολίτη, σοβιετικού πολίτη. Ευτυχώς κατέρευσε η δικτατορία της Ρουμανίας. Έγιναν συγκρούσεις βέβαια στους δρόμους ε, των Ρουμανικών πόλεων με την αστυνομία, αλλά η Ρουμανική Επανάσταση ήταν έμπνευση και σε γειτονικέ χώρες να αναλάβουν το πεπρωμένο στα χέρια τους. Ε, ευχαριστώ και συγχαρητήρια σε όλο το ρουμανικό έθνος. Σας ευχαριστούμε κύριε Τζαμπάτσκι. Το λόγο έχει ο κύριος Ζαχραντήλ για ένα λεπτό επίσης. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ επίκαιρος αυτός ο εορτασμός ε, της κατάρρευσης ε, του κομμουνιστικού καθεστώτος ε, στην Ρουμανία. Ήταν το τελευταίο δορυφορικό κράτος, το τελευταίο κατάλοιπο της κομμουνιστικής αυτοκρατορίας, το τελευταίο κομμουνιστικό καθεστώς που κατέρευσε. Και Μάλιστα ήταν και η πιο ε, βίαιη και αιματοβαμένη επανάσταση σε όλη τη διαδικασία της κατάρρευσης ε, της Σοβιετικής ηγεμονίας στην Ευρώπη, στην Ανατολική Ευρώπη. Εμείς ε, στην Τσεχία, στη τότε είχαμε τη χαρά της ε, ανέμακτης βελούδινης και η μετάβαση στο νέο δημοκρατικό σύστημα από το κομμουνιστικό καθεστώς ήταν πολύ ειρηνική ευτυχώ για μας. Πραγματικά όμως μας συγκλώνησαν, μας συντάραξαν οι τηλεπτικές εικόνες από τα γεγονότα στη Ρουμανία. Είχαμε την ε, εκτέλεση του Τσαουσέσκου όταν εμείς είχαμε ήδη μεταβατική κυβέρνηση και είχαμε ήδη ακολουθήσει το δρόμο προς τις ελεύθερες δημοκρατικές εκλογές. Πάντως, το τμήμα τη συνολική διαδικασία, είναι σημαντικό να θυμόμαστε αυτά τα γεγονότα και να τα εορτάζουμε και χαίρομαι γιατί υπερψηφίσαμε το σχετικό ψήφισμα. Σας ευχαριστώ κύριε Ζαχραντήλ. Υπήρχε ένα πρόβλημα με τη διερμηνία. Κύριε Χόρκιν, γιατί ζητήσετε το λόγο. Ναι, δεν άκουγα τίποτα. Ε, τώρα όμως ακούω τη διερμηνία. Ευχαριστούμε κύριε Γκέρκιν. Ο κύριος ε, Μπότος έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Και εγώ φυσικά υπερψήφισα το ψηφίσμα και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, που έπραξαν το ίδιο. Είναι πολύ σημαντική αυτή η στιγμή για τους συμπολίτε μου, για το λαό μου, για την ιστορία μας και είμαι πανευτυχής που ε, τονίσαμε τη σημασία αυτού του γεγονότος εδώ στο ιερό της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Τα γεγονότα του 1989 άλλαξαν ε, άρδιν την κατεύθυνση της Υπήρου, μας. Και χαίρομαι γι' αυτό και ευχαριστώ όλους ε, τους συνανθρώπους μας που έδωσαν τη ζωή τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Είναι σημαντικό λοιπόν να τιμούμε τη μνήμη τους και να στέλνουμε αυτό το μήνυμα από τον οίκο της Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου για την κατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα και να δώσω το λόγο στον στην Ντομινίκ Μπίλντε, συγγνώμη. Η κατάσταση των Ουιγούρων ε, ε, είναι κάτι ανάλογο με την κατάσταση των Ροίνγκια στη Βερμανία και τα ίδια μέτρα πρέπει να ληφθούν. Είναι φυσικό δικαίωμα ω ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δεν θα πρέπει όμω το ρεσπαστικό Ισλάμ να παρισφρεί στου κύκλου αυτή τη μικρή κινησική μειονότητα και να απειλεί την ταυτική ακαιρεότητα απέναντι σε έναν πάρα πολύ αγωνιστικό Ισλαμικό μιλιταρισμό. Έχουμε παραβιάσει θεμελιωδών δικαιωμάτων, Τη της ελευθερίας ε, συνείδησης. Πρέπει να διαπιστώσουμε όμως ότι υπάρχουν ε, ε, και κάποια κενά, τα οποία είναι πολύ παλιά στην Κίνα όμως. Παραδείγματο χάρη, χριστιανικό δόγμα από το 2017 δεν μπορεί να ασκηθεί με ελευθερία. Αυτό δεν το λαμβάνει κανείς υπόψη. Επίσης υπάρχουν πολλοί ε, παρενοχλήσεις ε, και δεν μπορούν ούτε τα κηρύγματα ε, να γίνουν όπως θα έπρεπε. Η αποφασιστικότητά μας είναι αυτή και η πυγμή μας είναι αυτή που θα πρέπει να υπερισχύσει απέναντι στην Κίνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπίλτελη Πρόεδρος. Προχωρούμε στις επεξηγήσεις ψήφου για την ε, κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στην Ικάρα. Ο συνάδελφος Γιάνν Ζάχραντιλ. Ευχαριστώ πολύ. Για μια ακόμη φορά έχουμε να κάνουμε το ίδιο θέμα και είναι πολύ θετικό που το συζητάμε και που εγκρίναμε και σχετικό ψήφισμα. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν μιλάμε για την Κεντρική Λατινική Αμερική, βλέπουμε να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμές. Συνάδελφοι της αριστερής πτέρυγας ε, αρέσκονται στο να ασκούν κριτική στα καθεστώτα ε, με τα οποία ε, δεν είναι ιδεολογικά στην ίδια θέση μαζί τους, όπως τη Χιλή ή τη Βραζιλία και την Κολομβία. Όταν όμως ε, πρόκειται για τη Βενεζουέλα ή την Κούβα ε, που είναι φιλικά προσκύμενες ε, τη Βολιβία ακόμα οι κυβερνήσεις. Ο πρόεδρος της Βολιβίας φυγαδεύτηκε, έφυγε από τη χώρα ή σε άλλες χώρες. Εκεί λιγότερο τους βλέπω πρόθυμους να ασκήσουν κριτική για την παρέμβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν πρέπει να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρος. Θα παρακαλέσω τον Πάτρικ Μπράιερ τώρα να πάρει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, οι πειρατές είμαστε υπέρ στο να λογοδοτήσουν ε, όσοι είναι δράστες ε, παραβίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Να υπάρχει και η ασυλία ε, για τον επικεφαλής ε, του κράτους. Και το ψήφισμα αυτό του Κοινοβουλίου για την Νικαράγουα δεν λαμβάνει υπόψη του ε, τα μέτρα αυτά, ιδίως εφόσον ζητεί κυρώσεις και κατά του Προέδρου της Νικαράγουα ε, και του ε, ασκούντος καθήκοντα αρχηγού κράτους αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό είχαμε ζητήσει και τμηματική ψηφοφορία, ειδικά για αυτό το κομμάτι. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος, και προχωρούμε. Βία καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν. Μάθιου Πάτεν, παρακαλώ. Um, Εγώ υπερψήφισα το ψήφισμα ε, που καταδικάζει την ε, βία καταστολή στο Ιράν και πραγματικά θρηνούμε τους θανάτους αλλά και τους πολιτικούς κρατούμενους ε, που πρέπει αμέσως να απελευθερωθούν. Αλλά θα πω το εξής. Τέτοιες χειρονομίες σαν αυτό το ψήφισμα δεν έχουν και τόσο νόημα. Οι συνάδελφοί μου συνήθως ε, ε, καταδικάζουν τη ΣΥΠΑ και τον πρόεδρο Τραμπ. Όμως η Αμερική είναι ο μόνος, το μόνο έθνος που έχει την ισχύ, τους πόρους και τις σχέσεις για να μας βοηθήσει να επιτύχουμε αυτό που επιθυμούμε να επιτύχουμε με αυτό το ψήφισμα. Προχωρώντας λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να σεβαστούν αυτόν που είναι ο μεγαλύτερο σύμμαχος της Ευρώπης εδώ και τόσα χρόνια και θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά, στο Ιράν πρέπει να ξεκινήσουμε στην Ουάσιγκτον. Ευχαριστώ πολύ και συνάδελφε Πάτεν και τώρα μπορώ να ανακοινώσω ότι κλείνει η συνεδρίαση μέχρι τις 3. Διακόπτεται μάλλον μέχρι τις 3. Για όσους δεν ξαναδούμε, καλές διακοπές, καλά Χριστούγεννα. Παναλαμβάνονται οι εργασίε ε, τη συνεδρίασης, ε, τα πρακτικά της συνεδρίασης και τα σχετικά κείμενα ε, είναι στη διάθεσή σα. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσει, θεωρούνται εγκεκριμένα τα κείμενα αυτά και προχωρούμε Σύμφωνα με την ουσία διάταξη, στην ανακοίνωση του αντιπροσώπου τον είπα για το εμπόριο σχετικά με την έρευνα δυνάμει τη ενότητα 301 για το φόρο ψηφιακών υπηρεσιών, να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε είτε με το συνηθισμένο τρόπο είτε με τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος να δηλώσετε συμμετοχή στη δικασία προσέξης προσοχής του Προέδρου ή μπλε κάρτα. Ξεκινούμε λοιπόν με το σημείο αυτό, με την δήλωση της Επιτροπής. Θα ακούσουμε τον Επίτροπο Χόγκαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έγιναν προτάσεις ε, ε, από την Κομισιόν για τη δίκαια φορολόγηση των εταιριών, να υπάρχει μια δίκαια φορολόγηση. Θέλουμε να βρεθεί μια μακροπρόθεσμη λύση που θα ορίζει και την έδρα, την εγκατάσταση, ώστε η ψηφιακή παρουσία ε, να εξασφαλίζει και τον σωστό συντελεστή για την εταιρική φορολόγηση. Την πρόταση αυτή της Κομισιόν πρέπει έναν χρόνο ε, τέλη Δεκεμβρίου την υποστήριξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατατέθηκε αυτή η πρόταση να αναμονή μια πιο συνολική λύση με στόχο να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενε πιέσει που ατομίζουν τα κράτη-μέλη για να λάβουν δράση επειδή υπάρχει διάβρωση της εταιρική φορολογικής τους βάση το χρόνο και για να υπάρχει δίκαιο ε, σύστημα. Θέλαμε να επιταχύνουμε και τη συζήτηση επίπεδο ΩΣΑ για να βρεθεί ένα συνολικό ε, πλαίσιο και για το φόρο ψηφιακών υπηρεσιών. Δυστυχώ ε, το Συμβούλιο δεν κατέληξε σε συμφωνία επί της προτάσεως της Κομισιόν αρχές του 2019. Η Γαλλία και κάποια άλλα κράτη-μέλη προχώρησαν να στην εκπόνηση ε, ε, εθνικών συστημάτων για το φόρο ψηφιακών υπηρεσιών και ξεκίνησε η έρευνα ε, της λεγόμενης ενότητας 301 είπα τον Ιούλιο του 2019 πρώτη φορά που είπα ερευνούν την περίπτωση αυτή χωρίς η Γαλλία να είναι όμως η πρώτη χώρα που είχε εγκρίνει ένα τέτοιο φόρο μετά από αυτά ο πρόεδρος Μαρκών ο πρόεδρος ε, στο G7 στον Πιαρίτσα αποφάσισαν ότι η Γαλλία θα συνεχίσει την εισπράξη αυτού του φόρου και θα επιστρέφεται αυτό ο φόρο σε αν υπάρχει διαφορά μεταξύ του γαλλικού φόρου και του συνολική λύσης τόσα. Παρά τη συμφωνία αυτή, συνέχισαν είπα, την έρευνα αυτή ε, και στις 2 Δεκεμβρίου του 2019 λένε ότι ο φόρος ψηφιακών υπηρεσιών της Γαλλίας είναι ε, δια, συνιστά δικαιωτική μεταχείριση, υπέρμετρο, συνιστά υπέρμετρη φορολόγηση και έτσι ε, ξεκίνησαν τη δικασία για τη θέσπιση και μονομερών μέτρων. Μόνο μία φορά έχει ξαναχρησιμοποιηθεί για την Κίνα, για θέμητες εμπορικές πρακτικές, για την οικονομία της ε, Κίνας που δεν θεωρείται οικονομία της αγοράς ε, για την αντιμετώπιση εμπορικών ε, διαφωνιών μόνο μέσω του ΠΟΕ είναι κανονικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα και έχουν χρησιμοποιήσει αυτέ τι διόδου, είπα, κατά το παρελθόν. Καλούμε λοιπόν ε, να μην ε, παραβιάσουν τι διεθνεί υποχρεώσει στο πλαίσιο του πολυμερού εμπορικού συστήματο ε, οι Αμερικανοί. Και η πρόεδρο Φοντερ είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δράσει και θα αντιδράσει κατά οποιοδήποτε μονομερού μέτρου εκτό του συστήματο του ΠΟΕ. Θα συνεχίσει δεν να προασπίζεται τα συμφέροντα των κρατών μελών αν ληφθούν μέτρα μονομερή σε βάρο του από κάποιο άλλο κράτο. Έχουμε τον κανονισμό Επιβολή επιβολής από Κοινοβούλιο και Συμβούλιο που στέλνει και ένα ηχηρό μήνυμα. Η Ένωση είναι έτοιμη να προστατεύσει και ε, τα συμφέροντα των χωρών της και το πολυμερι εμπορικό σύστημα. Επομένως, θα ανησυχούσε ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, η επιβολή τελικά ε, κυρώσεων, δασμών από του ΣΥΠΑ βάσει της έρευνας αυτής 301β θα είναι πρώτη φορά από το 1974 που χρησιμοποιείται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τότε που ουσιαστικά ιδρύθηκε ε, το 1995 ο ΠΟΕ είπα και εμείς ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει η συζητήση και ο διάλογος να είναι η διέξοδος και όχι η επιβολή μονομερών μέτρων. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε το διάλογο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επιτροπέ Χόγκαν. Η κυρία Βεντρέν έχει καταρχάς το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, είμαστε εδώ στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τελευταία συζήτηση του 2019. Μία συζήτηση που αντικατοπτρίζει την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε εδώ και πολλά χρόνια στο διεθνές εμπόριο. Το διεθνές εμπόριο είναι γνωστό τη σπάση ότι διανύει μια περίοδο αναταράξεων. Πολλά άλλαξαν. Η θέση τη κίνα, των ψηφιακών ε, τεχνολογιών. Αλλά καταφέραμε να προσαρμοστούμε στις αλλαγές. Όχι. Προσπαθούμε να ταχθούμε υπέρ ενό ισορροπημένου και βάση κανόνων διεθνού εμπορίου. Σήμερα εμεί οι Ευρωπαίοι υφιστάμεθα πιέσει και είμαστε στο στόχαστρο μια, για μια ακόμη φορά του Ντόναλτ Τραμπ. Μάλιστα αποφάσισε να επιβάλλει δασμούς εδώ και δύο χρόνια στο, στον ευρωπαϊκό χάλιβα και στο ευρωπαϊκό αλουμίνιο, κάτι που είναι παράνομο. Εμείς αντιδράσαμε με τι αποτελεσματικότητα όμως. Από τα μέσα Οκτωβρίου οι ευρωπαίοι παραγωγοί και αγρότες ε, υφίσταται πλέον τελωνιακούς δασμούς 25% μετά την υπόθεση Airbus Boeing και μάλιστα επέβαλε και 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ κυρώσεις. Και έκτοτε η κυβέρνηση του Τραμπ α, α, ανήγγειλε ότι θα επιβάλλει 100% δασμούς ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ε, α, ως αντίπεινα για τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών. Ε, εμείς ζητήσαμε να συμπεριληφθεί ε, αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη Ολομέλεια πριν την προθεσμία που έχουν οι Αμερικανοί τον Ιανουάριο. Γνωρίζω ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες μα. Τι μα προσάπτει ο Ντόναλτ Τραμπ. Θεωρεί ότι ο φόρο ψηφιακών υπηρεσιών συνιστά διακριτική μεταχείριση των Αμερικανικών εταιριών. Λάθο Είναι απλώ ε, ένα δίκαιο αντίτιμο που πρέπει να καταβάλουν οι ψηφιακέ εταιρείε. Άλλωστε, ζητούμε να βρεθεί μια παγκόσμια λύση στα πλαίσια του ΟΣΑ. Θα πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση και η διαπραγμάτευση ώστε να καταλήξουμε σε ένα δίκαιο ψηφιακό φόρο που θα εγγυάται ισότιμο ανταγωνισμό. Αυτή η επίθεση λοιπόν του Τραμπ ουσιαστικά στράφηκε κατά τη ε, γαλλική ε, σαμπάνια, του ροκφόρ, ε, του των καλλιντικών, των τσαντών, προσπαθεί να χτυπήσει τις ναυαρχίδες ουσιαστικά της ε, γαλλικής οικονομίας. Επίσης ανησυχητικό είναι ε, ότι θα επηρεαστούν με κάποιες πολυεθνικές, γαλλικές και ευρωπαϊκές, αλλά πιο πολύ θα ε, χτυπηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αγρότες μας. Τέτοιοι δασμοί θα είναι ολέθριοι για αυτούς και πληρώνουν αυτοί τα σπασμένα, οι αγρότες μας των εμπορικών μέτρων. Θα πρέπει λοιπόν σε περίπτωση που εφαρμοστούν τέτοιοι δασμοί να ληφθούν κάποια ε, μέτρα αποζημίωσης. Επιμένω στην ανάγκη διαλόγου μεταξύ δύο βασικών εταίρων. Θα πρέπει να πρετανεύσει ο διάλογο και να σταματήσει αυτή η διελκυστίδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ανέκαθεν ανοιχτή στη συζήτηση και ελπίζω να εισακουστούμε από τι ΗΠΑ. Γιατί μια τέτοια κλιμάκωση των ε, εμπορικών εντάσεων μόνο χαμένου θα έχει. Θα πρέπει να βρεθεί μια αμοιβαίω επωφελή λύση γιατί σε αντίθετη περίπτωση οι παραγωγοί και οι καταναλωτέ και των δύο πλευρών θα υποστούν τι ολέθριε συνέπειε μια τέτοια κλιμάκωση. Θα πρέπει επίση να διαφυλάξουμε την ενότητα των κρατών μελών. Αυτό είναι βασική μα αξία γιατί ε, η ενότητα είναι η βάση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το γονιδίωμά μα, το DNA μα Εν τη ενώση ισχύει. Θα πρέπει να το επαναλάβουμε και να το διατρανώσουμε. Η συζήτηση αυτή δείχνει πόσο επίγουσα είναι η ανάγκη. Θα πρέπει να ενισχύσουμε και να θωρακίσουμε την εμπορική μα πολιτική. Η δεμή θα πλήξουμε την ίδια μα την οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη ε, παγκοσμίω οικονομική δύναμη. Θα πρέπει λοιπόν να το διατρανώσουμε και να είμαστε πιο επιθετικοί στη συμπεριφορά μα. Και για να τελειώσω με τελευταία αναγγελία των ΗΠΑ, το μήνυμά μου σήμερα είναι σαφέ. Η κλιμάκωση των εντάσσεων που συνεχίζεται δεν είναι ούτε βιώσιμη ούτε λογική και θα πρέπει επιτέλου να τερματιστεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Βεντέν. Για τρία λεπτά το λόγο κύριο Τσαμπάτσκι. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Χόγκαν, συνάδελφε Βεντρέν, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι προνόμιο που συμμετέχω σήμερα σε αυτή την ε, επική και πολύ θερμή συζήτηση, ζωντανή συζήτηση ε, σήμερα στην Ολομέλεια. Είναι χαρακτηριστική η συμπεριφορά των Ευρωβουλευτών. 751 είμαστε και μόνο τέσσερις είστε σήμερα εδώ παρόντες ε, και θέλω να τιμήσω ο Πρόεδρο που είναι πολύ αυστηρός με το χρόνο ομιλίας. Υπάρχουν αρκετοί, μέλη εδώ, αρκετοί Ευρωβουλευτές εδώ για να παίξουν παίξουμε χαρτιά. Ε, είμαστε μόνο τέσσερις και... Επίσης αυτό που είναι ενδεικτικό είναι ότι οι θεατές ε, στα θεωρία είναι δέκα φορές περισσότεροι από μας τους ευρωβουλευτές. Αλλά εκείνοι είναι που επηρεάζονται περισσότερο, γιατί ο φόρος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα επηρεάσει όλες τις εφαρμογές και τις χρήσεις που κάνουν οι πολίτες, όλες τις συσκευές. Ε, που χρησιμοποιούν. Μπορείτε να δείτε πόσο ενδιαφερόμαστε για αυτή τη συζήτηση. Αλλά ας πούμε στην ουσία. Στις 10 Ιουλίου του 2019 ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΕΠΑ ξεκίνησε έρευνα όσον αφορά το γαλλικό φόρο ε, ε, ψηφιακών υπηρεσιών όπου προβλέπεται 3% φορολόγηση στα κύκλο εργασιών των εταιριών που λειτουργούν στο γαλλικό έδαφος. Οι εταιρείε που γεννούν παγκοσμίως 750 εκατομμύρια κέρδη και 25 εκατομμύρια κέρδη στην Γαλλία αφορά ο νόμος αυτός. Οι δηλώσεις ορισμένων Γάλλων ε, αξιωματούχων δείχνουν ότι αυτό ε, ο φόρος είναι δυσανάλογος και αδίκως επιβαρύνει τις αμερικανικές εταιρείε. Θα πρέπει ωστόσο να διατηρούμε αγαστές σχέσεις με τους γειτονές μας γιατί ε, οι αμοιβές ενέργειες ενέργειες από πλευράς ε, των ΗΠΑ δεν είναι προ το συμφέρον μα και μπορώ να παραθέσω τον εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στην ΗΠΑ και, στις ΗΠΑ και την Κίνα ω παράδειγμα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει κάτι τέτοιο γιατί πρόκειται για έναν από του πιο στενού εμπορικού μα εταίρου. Ε, θα εξακολουθήσω να μιλώ υπέρ του ελεύθερου εμπορίου. Είναι ο μόνο τρόπο για να εγγυηθούμε την εφημερία για όλου του πολίτε. Η Γαλλία δεν είναι ολόκληρη η Ευρώπη και ελπίζω πω άλλα κράτη-μέλη δεν θα, δεν θα ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. Επίση, θέλω να επιστήσω την προσοχή σε κάτι άλλο. Σε αυτή την αίθουσα συχνά ζητούμε εναρμόνιση του φορολογικού φόρτου ανάμεσα στα κράτη. Αυτά ε, στις εκκλήσεις κάνουν συνήθως οι κομμουνιστές συνάδελφοι και εμείς είμαστε αντίθετοι σε τέτοιες ε, προτάσεις. Η φορολογική πολιτική εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και εύχομαι καλές διακοπές σε όλους. Ευχαριστούμε κύριε Τσαμπάφσκι. Θα σας διορθώσω σε κάτι. Δεν είμαστε τέσσερις αλλά πέντε οι βουλευτές. Με ξεχάσατε μένα. Δεν με λάβατε υπόψη. Για τη διαδικασία προσέγγιση προσέγγιση δεν έχω κανέναν ε, που να έχει εγγραφεί στον κατάλογο, οπότε θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Χόγκαν. Α, κι όμω, να που υπάρχει. Η συνάδελφο έχει σηκώσει μπλε. Ναι, συγγνώμη. Άργησα λίγο να σηκώσω την κάρτα. Κυρίες και κύριοι, σε σχέση με τον συνάδελφο από το ECR θα συμφωνήσω ότι πραγματικά είναι πολύ απογοητευτικό επειδή γίνεται αυτή την ώρα η συζήτηση να μην είναι περισσότεροι βουλευτέ παρόντε στην αίθουσα. Τώρα έρχομαι σε εσά κύριε Χόγκαν. Θέλω να επικροτήσω και εσά και την ομάδα σα. Λίγες εβδομάδες μόνο έχετε αναλάβει τα νέα σας καθήκοντα, αλλά έχετε κάνει ήδη κάποια δουλειά ως εκπρόσωπος από την Ιρλανδία και από Midlands Northwest κυρίως. Θέλω να σας παρακαλέσω να συνεχίσετε να προωθείτε το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης, ιδίω σε ό,τι αφορά τα φορολικά, την ψηφιοποίηση και ελπίζω να θέσετε τα σχετικά ζητήματα σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς ε, με τους Αμερικανούς ομολόγους. Ε, Ποιαδήποτε υποστήριξη μπορείτε να έχετε από την Ιρλανδία θα την έχετε. Σας ευχαριστώ. Πρώτα σα ευχαριστώ πολύ συνάδελφε Walsh, λέει ο Τώρα έχετε το λόγο εσεί, κύριε Χόγκαν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τους ε, ευρωβουλευτές που επισήμαναν αυτό το ζήτημα και σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ε, για συνέχιση διαλόγου με τις ΗΠΑ για όλα τα εμπορικά θέματα και για το ψηφιακό φόρο φυσικά. Και θα, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι τον Ιανουάριο θα μεταβώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, αναζητώντας λύση σε αυτό το ακαθόδε ζήτημα. Και επ' ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς και την ομάδα σας, κύριε Πρόεδρε, το επιτελείο σας, ε, για την ε, πολύ αγαστή συνεργασία που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2019. Σας εύχομαι λοιπόν καλές γιορτές και ευτυχισμένο το νέο έτος 2020. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, κύριε και κύριοι. Εδώ ολοκληρώθηκαν οι σύνοδοι ολομέλειας του Κοινοβουλίου μας στο Στρασβούργο το 2019. Ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα ε, την Πέμπτη το απόγευμα. Ξέρουμε ότι οι περισσότεροι βουλευτές πρέπει να φύγουν ή έχουν ήδη φύγει. Αυτό μπορεί να μην το γνωρίζουν οι επισκέπτες μας αλλά έτσι είναι ο κύκλος ε, έτσι είναι οι εργασίες μας εδώ. Ε, πάντως ε, δεν πρέπει να ε, παραπονείστε διότι έχουν μαγνητοσκοπηθεί οι ομιλίες σας και οι ομιλίες σας μπορεί να παιχθούν στο διαδίκτυο και κανείς δεν θα ξέρει αν είναι την πέμπτα απόγευμα ή αν είναι την τετάρτο βράδυ και μπορεί να μην ξέρουν ακριβώς τι γίνεται και αν ήταν η λομέλη άδεια ή γεμάτη. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ ε, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και με ένα ευτυχισμένο νέο έτος. Εύχομαι σε όλους κάθε επιτυχία ε, και κάτι το οποίο δεν θα βλάπτει την πολιτική μας ε, πατρίδα, ελπίζω. Και θα τα ξαναπούμε. σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω τους βουλευτές ε, και τον Επίτροπο, αλλά και όλους ε, τους υπαλλήλους δεξιά, αριστερά, που κάθονται δηλαδή εξ ε, αριστερών και εκ δεξιών μου και τους διερμηνείς μας που ουσιαστικά είναι αυτοί που μας δίνουν φωνή διότι χωρίς τις διερμηνίες δεν θα καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας ε, και επειδή έχω και αυτή την προφορά εγώ που έχω, ε, ζητώ όλος ιδιαίτερο συγγνώμη από τους διερμηνείς. Κύριε Τζαμπάσκι, ε, είπατε ότι είμαι αυστηρός με, το χρόνο αγόρησης. τώρα δεν μπορώ να σας δώσω κανονικά το λόγο σε αυτό το σημείο με την πλεκάτα, αλλά θα σας το δώσω παρόλα αυτά. Του κουστόμου, Κοιτάξτε, εκτός και ε, ε, θα πρέπει να είστε πολύ αυστηρός με το χρόνο και παρακαλώ να συνεχίσετε να το κάνετε αυτό. Ε, και όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της Ολομέλειας και της, της ημερής συζητάξης, θα πρέπει να το σκεφτούμε πολύ καλά για το αν θα πρέπει καν να συνεδριάσουμε την Πέμπτη το απόγευμα. Είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει, να μας προβληματίσει. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εσάς, τον Επίτροπο, τους Διερμηνείς και σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και ευτυχία ευτυχισμένο Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τζαμπά, και τα πρακτικά αυτή της συνεδρία θα είναι διαθέσιμα προς έγκριση στην αρχή τη επόμενη συνόδου και τα ψηφίσματα ε, και τα ε, υπόλοιπα κείμενα θα ε, υποβληθούν σε όσους πρέπει. Σας εύχομαι όλους καλές γιορτές. Λήξη της συνεδρίασης.